Colleghi, buonasera. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Ξεκινάμε τα τις εργασίες της απογευματινής συνεδριάσεως σχετικά με τις ανακοινώσεις από την έκβαση της συνεδριάσεως των συντονιστών έχω να σας πω ότι σχετικά με την σημερινή ημερήσια διάταξη οι ε, συντονιστές συμφώνησαν στο πρώτο σημείο εις ε, την ε, την αποστολή για τον Οκτώβριο στην Πολωνία και θα ανακαθοριστεί η σύσταση της αποστολής η οποία θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 24 ώρων για να ενημερώσουμε αρμοδίως την Προεδρία η οποία θα συντονίσει την οργάνωση. Συμφωνήσαμε ότι σχετικά με την ψηφοφορία για το αέριο αποσκιστόλιο για τις 9 Οκτωβρίου υπάρχει ένας καθορισμός του προγράμματος σχετικά με την συμμετοχή των πολιτών που έχουν προσυπογράψει την αναφορά και των ομιλητών που θα δώσουν τεχνική γνωμοδότηση. Τα σημεία 4 και 5 ανεβλήθησαν κατόπιν αιτήσεων του ΕΛΚ που τα είχε υποβάλει. Όσον αφορά το θέμα της κοινή ε, ε, συμφωνίας της, ε, της κοινής συνεδριάσεως της Επιτροπής Αναφορών με, την, με μια άλλη επιτροπή αποφάσισε να γίνει τον Ιανουάριο του 2013 και έχει αποφασιστεί όπως αποφασίστηκε να συζητήσουμε εκτός του σημείου 19 τις ε, ε, αναφορές και ε, για τις τεχνικές ανακοινώσεις αποφασίστηκε ότι θα περιμένουμε και την παρουσία του, της, συνήθου, της συναδέλφου Τουργκάη και να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά της ε, με ε, την ε, υποτινέρεση ότι είναι αποδεκτή. Δεν λήφθηκαν άλλες αποφάσεις από τους συντονιστές και αν δεν υπάρχουν επεμβάσεις για χρόνο ομιλίας και παρεμβάσεις θα περάσω στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως Έχουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως την αναφορά 771-2012 του, του κυρίου Μαουρίτσιο Λαντσελότη. Πρόκειται για μία μεμονωμένη αναφορά υπάρχουν εκπρόσωποι της ε, τοπικής κοινωνίας οι οποίοι ζήτησαν να λάβουν το λόγο και ε, αποφασίσαμε ότι επειδή υπάρχει περιορισμένος χρόνος ε, ομιλίας θα δώσω καταρχήν το λόγο στον υπογράφοντα τον κύριο Μαουρίσιο ο Λαντσελότο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που δεχθήκατε να συζητήσουμε μαζί την αναφορά που καταθέτουν 400.000 κάτοικοι της Βόρειας Ρώμης που εδώ και δύο χρόνια προσπαθούν να προασπίσουν την υγεία τους και τις συνθήκες υγιεινής. Από τότε που η Ευρώπη προχώρησε στην προσφυγή παραλήψη για την ελληματική διαχείριση των αποβλήτων στο Λάτιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ήδη από τις 6 Ιουλίου του, του 12, ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα αυτά στη Ρώμη προσπάθησε να προχωρήσει στη λήψη μέτρων. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι προς στιγμήν η συγκεκριμένη περιοχή δεν προορίζεται για μια νέα χωματερή, είναι κάτι η μαλαγκρότα, δεν είναι κάτι το οποίο μας καλύπτει. Μιλάμε για την ε, Ιταλική κομπίνα ουσιαστικά, είναι μια κομπίνα η οποία τροφοδοτεί τις μαφίες. Τα θεσμικά όργανα της Ιταλίας απέδειξαν την ικανότητά τους να διαχειριστούν τα απόβλητα σύμφωνα με τις ε, καθορισμένες προτεραιότητες της Οδηγίας 98-2008 αντιστρέφοντας την πυραμίδα μετα, ε, μεταχείρισης των αποβλήτων. Αυτό κατέστησε τη Μαλαγκρότα την πιο μεγάλη χωματερή της Ευρώπης και το κλείσιμό της οδήγησε το Λάτιο σε μια περιβαλλοντική καταστροφή ε, αναγκάζοντας τον προεδρεύοντα της περιοχής του Λάτιου να ορίσει έναν έκτακτο επίτροπο, ο οποίος αποφάσισε να ανοίξει νέες χωματορές παρεκκλίνοντας από τις οδηγίες και όχι να βελτιώσει την κατάσταση. Εντοπίστηκαν 7 νέοι τόποι στην περιοχή του Λάτιου. Η μελέτη αυτή έγινε χωρίς να γίνουν τεχνικές έρευνες και χωρίς σε καμία περίπτωση να ληφθεί υπόψη η οδηγία αποβλήτων και οι βέλτιστες τεχνικές πρακτικές διαθέσιμες. Η επιλογή ε, του να δημιουργηθούν νέες χωματερές στην περιοχή του Όλμο και στο Κουάντρο Άλτο και στην περιοχή του Ριάνο δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στους κατοίκους λόγω της μη διαβούλευσης και ε, λόγω της μη συμμετοχής των τοπικών αρχόντων. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιλογή αυτή ήταν καθαρά πολιτική, δηλαδή εκλογική. Ε, οι χωματερές δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα σωστό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες. Τα προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να έχουν σαν, στόχο, έχουν σαν στόχο τη μείωση των αποβλήτων και οι χωματερές δεν θεωρούνται ε, σωστά, σωστοί τόποι εναπόθεσης και ήδη έχει προχωρήσει το θέμα και στη Μαραγκρότα ε, ε, υπήρξε αγορά ε, των συγκεκριμένων εδαφών. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν οι κάτοικοι του Ριάνο προσπαθούν να προστατεύσουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Δημιούργησαν πολλές τοπικές επιτροπές οι οποίες κάθε μία από την πλευρά της συμμετέχουν στην επιλογή κατά της επιλογής του κάντρο Άλτο και του Πλάντε Λόλμο. Οι μελέτες έχουν δείξει, οι τεχνικές, ότι ο εντοπισμός του Quadro Alto και του Plan del είναι θα έλεγα καρπός παραλήψεων, λανθασμένων διαπιστώσεων ε, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις Οικομαφίες όπως επίσης και από την Επιτροπή που ασχολείται με θέματα ποινική δικαιοσύνης. το περιβάλλον το οποίο έχουν επιλέξει είναι η Παρθένο θα λέγαμε άγριο και προστατεύεται από την UNESCO ε, σαν ε, κληρονομιά της ανθρωπότητας και της περιοχής του Ριάνο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στα παιδιά μας από μια απαράδεκτη μειοπική πολιτική που καταστρέφει σαν καρκίνος τον ιστό, τον γεωγραφικό και τον κοινωνικό της περιοχής, γιατί οι περιοχές αυτές είναι περιοχές πνεύμονες για τις πόλεις. Εδώ βλέπετε το Πλάν βλέπετε δηλαδή την Τοσκάνη μέσα στη Ρώμη. Ε, δυστυχώς όμως ε, ε, οι επιλογές που έγιναν έχουν εν πολλής ακολουθήσει πάρα πολλές αλλαγές χρήσης των εδαφών. Πάνω σε τέτοια εδάφη οικοδομήθηκε η Ρώμη και οι περιοχές γύρω από τη Ρώμη. Έχουμε πάρα πολλά ήδη δώσει στον τομέα του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να συνεχιστεί η καταστροφή. Εδώ βλέπετε με κόκκινο την περιοχή του Λόλμο. Ε, Δεν έγιναν ε, μετρήσεις ε, παρά μόνο οι αποστάσεις σύμφωνα με το χάρτη Google από τις αστικές περιοχές. 750, 695 μέτρα από το Λόλμο και ανάμεσα στο Λόλμο και στο Κουάντρο Άρτο. Από το ιστορικό κέντρο του Ριάνο η απόσταση είναι 1400 με 2200 ε, νομίζω ότι οι αναλύσεις οι δικές μας δείχνουν ότι οι πολίτες ε, του Ριάνο θα έχουν προβλήματα με άσχημες μυρωδιές ε, στο 65% του χρόνου, δηλαδή 235 ημέρες το χρόνο. Ακόμα και κτίρια που απαιτούν ειδική προσοχή όπως σχολεία, οικοτροφία, γυροκομεία κτλ είναι σε αποστάσεις οι οποίες είναι σαφώς μικρότερες από αυτές που προβλέπονται. Για τη σωστή ανάλυση του Σάτινγκ δόθηκαν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι ξεπερασμένες εδώ και 10 χρόνια. Οι τεχνικές μελέτες των πολιτών του Ριάνο έδειξαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά γεωλογικά επικίνδυνα στοιχεία επικαλύψεις και υδρογεωλογικές βλάβες στο σύνολο της περιοχής, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από μελέτες ε, καθηγητών πανεπιστημίων και από το Ινστιτούτο Έρευνας των Υδάτων. Ο οιδάτινη πόροι της περιοχής ε, είναι ιδιαίτερα δραστήριη στην περιοχή του, ε, του, Πλάντε Λόλμο. Καλύπτεται η περιοχή από αργυλικά εδάφη και στην περιοχή του Κουάντρο Άλτο αλλά και του Πιάντελόλμο σε καμία περίπτωση δεν ελήφθησαν υπόψη οι προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής τη της περιοχής. Το Πλάντελόλμο υπάρχει μια ρωμαϊκή νεκρόπολη και ένας πύργος μεσαιωνικός. Οι Ιταλικές αρχές ε, ε, εντόπισαν με την μελέτη αυτή χωρίς ε, καθόλου θεμελιωμένη εννέα νέους τόπους για την εναπόθεση των αποβλήτων. Εμείς ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρέμβει για να προστατεύσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την κοιλάδα του Τίβερη, για να καταδικάσει το Ιταλικό κράτος και την περιφέρεια του Λάτιου για την επιλογή αυτών των δύο τόπων, του Κουάντρο Άλτο και του Πλάντε Λόλμο, που είναι ασύμβατοι για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα για να ζητηθεί η αποζημίωση προς τους τοπικούς πληθυσμούς σε επίπεδο τεχνικό, νομικό και οικονομικό. Και τέλος, ε, ζητάμε η, περιοχή, αναφορά αυτή να δοθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει επίσης συμμετοχή στις ακροάσεις του αρμόδιου έκτακτου επιτρόπου των τοπικών και περιφερειακών Ιταλικών αρχών. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο για την επόμενη παρέμβαση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε προσκαλέσει και τον έκτακτο επίτροπο, τον κύριο Γκοφρέντο Σορτήλε, ο οποίος μας διαβίβασε ότι δεν μπορεί να παραστεί και μας απέστειλε ένα σημείωμα στο οποίο μιλάω σε πρόσωπο της Επιτροπής και λέει ότι θα πρέπει ε, προς το παρόν να θεωρηθεί ότι ε, έληξε το θέμα, διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά η περιοχή του πιάντε Λόλμο, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ λύσεις και έχει ε, πει ότι θα γίνει μια επόμενη συνάντηση, κατά πάσα πιθανότητα στη διερευνητική επίσκεψη που θα γίνει το φθινόπωρο από την Επιτροπή μας. Να δώσω τώρα απευθείας το λόγο στον κύριο Πιέτρο Ντομένικο Μπερτούτσι, ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή Πολιτών ε, Νόντις Κάρικα. Ε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Αναφορών, διότι μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ παρόντες σήμερα. Εκπροσωπώ την τεχνική ομάδα της Επιτροπής ε, Ριάνο Νόντις Κάρικα και της Επιτροπής Τζέρο ε, Ριάνο, μηδενικά απόβλητα στο Ριάνο και Ριάνο Νοντισκάρικα. Και είμαστε εδώ όχι μόνο γιατί δεν θέλουμε απόβλητα στην περιοχή του Ριάνου, αλλά για να επαναλάμβουν ότι είμαστε κατά τη κατασκευή ε, μεγάλων χώρων διάθεσης αποβλήτων, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε συνεχή ε, ανανέωση των αποβλήτων. Καταρχά, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μα, θα θέλαμε να επαναλάβουμε κάποια αιτήματα τα οποία θα θέλαμε να απευθύνουμε στην Επιτροπή σα και επίση να σα δώσουμε και κάποιε τεχνικέ ενδείξει που υποστηρίζουν τα αιτήματά μα. Καταρχάς, τις περιοχές ε, Κουάντρο Άλτο και Πιάντε Λόλμο, στην προκατακτική ανάλυση που έγινε για να βρεθεί ε, ε, αν είναι κατάλληλες για ε, χώρους διάθεσης αποβλήτων, διαπιστώνουμε ότι είναι πανομοιότυποι από, με άλλα προγράμματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν και αυτά τα προγράμματα είχαν απορριφθεί και από το Δήμο του Ριάνο και από την Ομαρχία, διότι θεωρούμε ότι αντιβαίνουν στα ε, τοπικά, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα. Καταρχάς, οι περιοχές αυτές είναι αντίθετες με τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο του 2007 για την ανάπτυξη της περιοχής ε, και λέγεται ότι σε όλη την ενδιαφερόμενη περιοχή απαγορεύεται ρητά, προτείνεται ρητά να μην υπάρχουν χώροι ε, διάθεσης αποβλήτων. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο της Ρώμης και η εισαγγελία μίλησαν με την Ένωση Περιβάλλον και Ζωή και Λέγεται ότι το θέμα της διάθεσης των αποβλήτων είναι μεν αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να γίνει βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αρκετοί κανόνες οι οποίοι δεν έγιναν σεβαστοί. Για παράδειγμα, η Οδηγία 1999-31 η οποία μεταφέρθηκε με, την, ε, ε, με το Προεδρικό Διάταγμα 36-2007 της Ταλικής Κυβέρνησης που λέει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η απόσταση από κατοκιμένες περιοχές, οι γεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, η οδηγία 85 85-337, η οποία αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η 2001-42 για την στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Ε, η σύμβαση του Άρχους ε, για τις δημόσιες συμβάσεις, ε, για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, συγγνώμη, και ε, για το γεγονός ότι ε, όλα αυτά θα είναι επιζήμια για την οικονομία και την εικόνα μιας ολόκληρης κοινότητας. Όλα αυτά λοιπόν αντιβαίνουν σε όλη αυτή την νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ε, και να πούμε ότι η προκαταρκτική ε, ανάλυση δεν είναι έγκυρη και οι περιοχές του Πιάντε Λόλμο και του Ριάνο δεν είναι κατάλληλε κατάλληλες περιοχές. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή σας να δραστηριοποιηθεί στα όσα την αφορούν φυσικά και την αρμοδιότητά της, καταρχάς ώστε να διευκρινιστεί ότι η προκαταρκτική ανάλυση αντιβαίνει με την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ότι στην περιοχή του Λάτιο και σε άλλες ε, σε άλλους ε, ε, θεσμικά όργανα, όπως για παράδειγμα στον Επίτροπο της Κυβέρνησης ή στις αρμόδιες αρχές, δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοιες αναλύσεις. Επίσης, ο αρμόδιος έκτακτος επίτροπος, ο κύριος Σωτήλη, θα πρέπει να κυρώσει την 2011 2086-25, βάσει της οποίας η περιοχή του Πιάντελάλτο θεωρείται κατάλληλη για χώρο διάθεσης αποβλήτων, όπως προέβλεψε ο προηγούμενος Επίτροπης. Επίσης, ο κύριος Σωτήλο θα πρέπει να κυρώσει το τμήμα του διατάγματος του 2012-56, ε, βάσει του οποίου η περιοχή αυτή είναι ιδανική για προσωρινή διάθεση αποβλήτων. Και επίσης, επειδή αυτές οι δύο περιοχές δεν είναι η κατάλληλη, θα πρέπει η Επιτροπή σας, εφόσον το αποφασίσει, να δηλώσει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν αυτές ε, οι περιοχές χώροι διάθεση αποβλήτων. Εμείς σας ζητούμε να προστατεύσετε την υγεία, το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα τηρήσετε την ένωμη τάξη. Ολοκληρώνω. Για τις ε, περιοχές αυτές μίλησαν οι αρχές ε, για τη λεκάνη του Τίβερη η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, της Βουλής, ε, το Τμήμα ε, Προστασίας του Περιβάλλοντος της περιοχής της Ρώμης, το Συμβούλιο της Ρώμης, το Συμβούλιο του Δήμου της Ρώμης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Ριάνου, 18 Δήμοι της Κοιλάδας του Τίβερη, καθώς επίσης και ο Δήμος της Ρώμης και 150.000 περίπου πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Δήμαρχο του Ριάνο, την κυρία Ριτσέλη, για να κλείσει τις παρεμβάσεις. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Νομίζω ότι επαρκώς υπογραμμίστηκε όλο το τεχνικό και πληροφοριακό κομμάτι γύρω από το σχέδιο αυτό των χωματερών στα εδάφη μας. Εγώ εδώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της πόλης μου και όλων των γειτονικών μικρών πόλεων. Το Ριάνο ανήκει σε μια ομάδα πόλεων οι οποίες εντάσσονται στην κοιλάδα του Τίβερη και συνορεύουν με την πόλη της Ρώμης. Είμαστε, θα έλεγα, ο τελευταίος πράσινος πνεύμονας της πρωτεύουσα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μιας και ακούστηκαν τα περισσότερα, το πώς η περιοχή μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μιας χωματερής στην περιφέρειά της, χωρίς να διαβουλευτεί κανείς με αυτήν. Εμείς, αν θέλετε, μας ανακοινώθηκε απλά μέσω του τύπου μάλιστα βασικά ότι το Ριάνο και το Κουάντρο Άλτο γενικότερα έχει επιλογή σαν μέρος υποδοχής αποβλήτων. Και το ίδιο συνέβη και με το Πλάν Τελόλμο. Βέβαια ένα χρόνο μετά, γιατί για μας εδώ και ένα χρόνο ασχολούμεθα με το θέμα αυτό, δημιουργήθηκαν επιτροπές, ομάδες διαμαρτυρίας για να καταπολεμήσουμε αυτές τις επιλογές οι οποίες έγιναν στο όνομα πίου Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε. Πρέπει να υπογραμμίσουμε βέβαια τις ζημίες τις οποίες, οι οποίες προκαλούνται στην περιοχή μας και στις γειτονικές μικρές πόλεις. Στο Ριάνο δεν υπάρχει μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Ίσως ε, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι των ε, οικοδομών, των κατασκευών και καταλαβαίνετε τι συνέπειες για αυτή τη δραστηριότητα υπάρχουν. Η βλάβη λοιπόν την οποία υφιστάμεθα εδώ και ένα χρόνο γιατί έχουμε χαρακτηριστεί σαν η πόλη των αποβλήτων. Ποιος θα μας αποζομιώσει, ακόμα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Ιταλικής Βουλής εδώ και λίγες μέρες είχαν κατατεθεί οι εργασίες εκεί που έγιναν όλο αυτό το χρόνο, συνειδητοποίησε το τι ε, έχει συμβεί Εμείς δεν θέλουμε τα απόβλητα, όχι γιατί δεν μας αρέσουν τα απόβλητα, αλλά γιατί η επιλογή στη συγκεκριμένη περιοχή έγινε με εντελώς λανθασμένο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν στην επόμενη φορά που θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Ρώμη και να καλέσω και τη δική σας Επιτροπή να έρθει οι ε, εκπρόσωποι της Επιτροπής της Βουλής μας είδαν επιτόπου τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σαν μια κακή ταινία όλη αυτή η ιστορία. Εδώ και ένα χρόνο ζούμε ένα κακό όνειρο με λίγα λόγια. Ευχαριστώ τη Δήμαρχο του Ριάνο. Λοιπόν, Ακούσαμε τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται και στις αναφορές. Δόθηκαν πληροφορίες από τους πολίτες. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Μαγκανάρο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε για την κατάσταση τη διαχείριση των απευλάτων στην περιοχή του Λάτιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά το ζήτημα εδώ και αρκετά χρόνια πλέον Υπάρχει μια διαδικασία επί παραβάση εν εξελίξη αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση της χωματερής της Μαλαγκρότα στην περιοχή, στα πλαίσια συγγνώμη, της οποίας ε, τον ε, ε, Ιούνιο, στις 12 Ιουνίου απεστήλει αιτιολογημένη γνωμοδότηση που ζητήθηκε στην οποία ζητήθηκε από τις Ιταλικές Αρχές να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται σωστή διαχείριση της περιοχής της Μαλαγκρότα Ξεκίνησαν και άλλες έρευνες στη συνέχεια που αφορούν και πάλι τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή του Λάτιο. Μία αφορά τη διαχείριση για την περίοδο μετά τη Μολαγκρότα, διότι οι Ιταλικές αρχές ανακοίνησαν την πρόθεσή τους να κλείσει ο χιτά στη Μολαγκρότα. Η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις για το πώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την περίοδο μετά το κλείσιμο της Μαλαγκρότα, τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ιταλικές αρχές ε, για τα όσα έχουν ήδη εγκριθεί, προκειμένου να γίνει κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή του Λάτιο. Αυτή τη στιγμή θα έχει κλείσει ο Χιτά στη Μαλαγκρότα σκοπεύουν να αυξήσουν την διαφοροποιημένη συλλογή, την κομποστοποίηση, ε, την ανακύκλωση, να υποχρεώνουν τον κόσμο να κάνει διάθεση αποβλήτων με συγκεκριμένο τρόπο. Τι σκοπεύουν να κάνουν. Επίση, κατόπιν καταγγελία που δεχτήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητήθηκαν και κάποιε διευκρινήσει από τι Ιταλικέ Αρχέ για την εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε θέματα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι ο έκτακτο επίτροπο, ο οποίο ορίστηκε προκειμένου να διαχειριστεί διαχειριστεί το κατεπήγον ζήτημα των αποβλήτων έχει την εξουσία να παρεκκλίνει από κάποιους κανόνες, ιδίως σε θέματα ε, διαβούλευσης ε, του κοινού και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συγκεκριμένα έργα. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμησε στις Ιταλικές Αρχές ότι αυτές οι παρεκκλήσεις δεν συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δηλαδή, εάν προκύψει ότι οι Ιταλικές Αρχές έχουν δώσει έγκριση για ένα σχέδιο ε, χώρων υγειονομική ταφή αποβλήτων χωρί να έχει ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει γίνει και διαβούλευση με το κοινό, αυτό αποτελεί παραβίαση του κοινωτικού δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και να δώσω το λόγο στην κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ τους πολίτες, τους αναφερομένους και εκπροσώπους των τοπικών αρχών, να καλωσορίσω την Δήμαρχο που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο Δήμο αλλά και τις άλλες κοινότητες της περιοχής που συνολικά φτάνουν σχεδόν τους 400.000, είναι πολύ μεγάλη αστική περιοχή. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Αναφορών, την Πρόεδρο Ματσόνη, γιατί θέλησε να επιταχύνει τη διαδικασία για την ακρόαση αυτή. Θα κάνω κάποια σχόλια γιατί εσείς τα είπατε όλα με πληρέστατο τρόπο. Όλοι αναφέρθηκαν σε έναν κατάλογο εγγράφων και επισήμων εντύπων, πέρα από τη δυστημία που νιώθει λοιπόν ο τοπικός πληθυσμός, πέρα από τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να μην θεωρηθούν υποκειμενικά, απαιτείται να υπάρξει σεβασμός για τα λεγόμενα αντικειμενικά δεδομένα, δηλαδή τα μετρήσιμα, αξιολογήσιμα και μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Εσείς έχετε εδώ συγκεντρώσει πάρα πολλά τεκμήρια από αρχές υπηρεσίες, ενώσεις που εξέδωσαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, που εξέθεσαν κάτι παραπάνω από ανησυχίες, που είπαν ξεκάθαρα ότι οι περιοχές αυτές είναι ακατάλληλες για μια ολόκληρη σειρά από λόγους ε, είτε για τους υδάτινους πόρους, ε, είτε για την κατάσταση των εδαφών, είτε για μία ε, κατάσταση ευαίσθητη υδρογεολογικά, ακόμα και ο Δήμος της Ρώμης, οι κοινότητες συνολικά της περιοχής του Τίβερη, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τις τελευταίες σου αποφάσεις και άλλοι δήμαρχοι επίσης μας θύμισαν και μια πολύ πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον γύρω από το θέμα των αποβλήτων. Υπάρχει λοιπόν αντικειμενικά θα έλεγα μια σωστή τεκμηρίωση πέραν των μεμονωμένων θέσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτές υποκειμενικές. Είναι σαφές ότι είναι πολύ θετική η επιστολή που έστειλε ο αρμόδιος έκτακτος επίτροπος για τα απόβλητα της περιοχής, ο οποίος λέγει ότι η απουσία του οφείλεται στο ότι η προσπάθεια εντοπισμού της συγκεκριμένης ε, περιοχής του Πλάντελόλμο πρέπει να θεωρηθεί ξεπερασμένη. Προς στιγμήν βέβαια διευκρινίζει. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι οι τοπικές αρχές και οι εκπρόσωποι ακριβώς όλων των περιοχών αυτών θα πρέπει να απαιτήσουν περισσότερη διαφάνεια. Εάν η περιοχή αυτή είναι ακατάλληλη για μία ολόκληρη σειρά λόγων, τότε θα πρέπει να διαγραφεί από αυτόν τον δυνητικό κατάλογο υποδοχής. Θα πρέπει να διαγραφεί. Και σε αυτή την περίπτωση θα κλείσει η υπόθεση. Συμπερασματικά θα ήθελα να προσθέσω, επανερχόμενος σε αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ότι η Ιταλία θα πρέπει να σεβαστεί τους κοινοτικούς κανονισμούς, θα πρέπει να σεβαστεί τις οδηγίες της σχετικές με το περιβάλλον και σεβόμενη η Ιταλία τις ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να φέρει εις πέρα στις υποχρεώσεις που έχει που υποχρεώνεται δηλαδή η χώρα και οι τοπικές αρχές να ενημερώνουν σωστά και να διαβουλεύονται με, τις, με τους κατοίκους και τις περιοχές οι οποίες συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Πρόεδρε, ευχαριστώ λοιπόν για την ενημέρωση. Ίσως θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να πάμε στο Ριάνο για να εκτιμήσουμε επιτόπου και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο τοπίου στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης η οποία προβλέπεται τον μήνα Οκτώβριο στη Ρώμη. Είναι επίγον να καταλήξουμε σε μια κάποια απόφαση και το επίγον είναι θα έλεγα εξηγείται από το ότι υπάρχουν εργολάβοι και επιχειρηματίες των οποίων οι εργασίες έχουν ουσιαστικά διακοπεί. Ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. Το λόγο θα πάρει ο κύριος Αντωνιώτση. Παρακαλώ ε, να μην μακρηγορήσετε. Πόσα λεπτά κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω ότι Αντιμετωπίσαμε τα πράγματα με επαγγελματικότητα και αποτελεσματικότητα. Ούτω ή άλλω ε, η Επιτροπή σα είναι καθήλυνα αρμόδια. Συγχαίρω και τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι επιτάχυναν τι διαδικασίε. Διότι είχαμε τους πολίτες που έξω τον κόδωνα του κινδύνου και ήταν κοινωνικό το πρόβλημα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που λάβατε υπόψη σας και τους κατόκους της περιοχής. Η Επιτροπή ασχολήθηκε πρόσφατα με την περιοχή του Κορκόλε, μια ε, άλλη κοινότητα, κοντά σε μια άλλη περιοχή προστατευόμενη από την UNESCO στη Βίλα του Ανδριανού. Η συζήτηση που έγινε τότε η οποία οδήγησε και σε πάρα πολλές επικρίσεις επειδή επελέγει συγκεκριμένη ε, περιοχή, τώρα επαναλαμβάνεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Πιάντελόλμο. Με μία διαφορά. Στην περιοχή του Πιάντελόλμο δεν είναι μόνο αρχαιολογικά μνημεία, δεν υπάρχουν μόνο υλικά αγαθά, υπάρχουν και πολίτες, ε, άνθρωποι, οικογένειες ε, και τα σπίτια τους φυσικά οι λόγοι για τους οποίους ε, το Πιάντε Λόλμο και το Κουάντρο Άλτο θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο των ε, περιοχών που θα έχουν ε, χώρους διάθεση απευλήτου είναι σαφής. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα το οποίο είναι πιο σημαντικό. Το γεγονός ότι δίνεται η εντύπωση ότι προχωρούμε και κάθε φορά έχουμε μια κληροτίδα και βγάζουμε, ε, επιλέγουμε μια περιοχή και όχι μια άλλη. Από το κορκόλε που ήταν λανθασμένο, φτάνουμε στο πιάντελόλμο που ήταν ακόμα πιο λανθασμένο και ποιο ξέρει που θα καταλήξουμε. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο θα ήθελα να θίξω σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας και σας ευχαριστώ, είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Είναι αδιανόητο να μην γνωρίζουμε ποια είναι η επιστημονική μέθοδος, όχι η τυχαία μέθοδος ή η πολιτική μέθοδος ή οποιαδήποτε άλλη φύσεως για την οποία αναζητούμε μια εναλλακτική λύση όταν θα κλείσει η, μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης, που είναι η χωματερή της Μαλαγκρότα. Το λέω γιατί υπάρχουν και μέλη εδώ στην Επιτροπή που δεν είναι Ιταλοί, που καλό είναι να γνωρίζουν και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Ζητούμε να επανεξεταστεί η μέθοδος μέσω της, οποίας, ε, μέσω της οποίας καταλήγουμε στη συγκεκριμένη επιλογή κάθε φορά. Και υπάρχει και κάτι το οποίο εξακολουθεί να με ανησυχεί. Στην ε, επιστολή που απέστειλε ο Επίτροπος ε, Σωτήλε, όπως μας διάβασε και η κυρία Αντζελίλη, εγώ δεν καθησυχάζομαι καθόλου, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κατάσταση της μελέτης και λέει ότι στη μελέτη ε, έχουμε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Το θέμα είναι ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικέ λύσεις. Ε, και το θέμα είναι ότι όλη η περιοχή της ε, ε Βόρειας Ρώμης, Βόρεια της Ρώμης μάλλον, έχει περίπου 400.000 κατοίκους και όλοι αυτοί θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Και το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ραγδαία διαδικασία χωρί να λάβει υπόψη της, ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εθνική, την περιφερειακή νομοθεσία, την περιβαλλοντική νομοθεσία, το σύνολο δηλαδή των κανόνων που προηγουμένω μα είπε ο πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό λοιπόν είναι το ευρύτερο ζήτημα εντό του οποίου τοποθετείται και η προστασία μια περιοχή, όπω είναι το Ριάνο. Το Ριάνο είναι και πανέμορφο συν τη άλλη. Ε, έχει φυσικό κάλος ε, από τα πιο ωραία της, ε, της Ιταλίας και δεν μπορεί κανείς να φανταστείς πώς καταλήξαμε χωρίς καμία επιστημονική έρευνα, χωρίς καμία ενεργοποίηση διαδικασιών να θεωρήσουμε ή να διανοηθούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια οικολογική καταστροφή και περιβαλλοντική ε, καταστροφή με τη δημιουργία ενός χώρου διάθεσης αποβλήτων για μια τόσο μεγάλη περιοχή όπως είναι η περιοχή της Ρώμης. Ε, θα θέλαμε να συνεχίσουμε να προσέχουμε το ζήτημα αυτό, όχι μόνο για την περιοχή του Κορκόλε και του Ριάνου, αλλά το σύνολο του ζητήματος, το όλο ζήτημα, Περιμένουμε και την επίσημη επίσκεψη η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο και θα ήθελα και εγώ να ζητήσω όπως και η συνάδελφος Αντζελίλη να μπορέσουμε να μεταβούμε επιτόπου ώστε οι επίτροποι να αντιληφθούν ότι τα μέλη της Επιτροπής μάλλον να αντιληφθούν ότι ε, αν μη τι άλλο, αν όχι προσβολή, είναι σίγουρα σχιζοφρενής η διαδικασία που ακολουθείτε. να πω ε, και πάλι ότι τα όσα μας λέει ο κύριος Σωτήλε δεν μας καθησυχάζουν καθόλου, ίσα ίσα μας ανησυχούν περισσότερο, διότι είχαμε και την προηγούμενη διαδικασία και την προηγούμενη δήλωση. Ο κύριος Σωτήλε μας είχε πει ότι η λύση του Ριάννου ήταν η οριστική απόφαση εκτός και αν ε, οι περαιτέρω επαληθεύσεις που γίνονται ε, αποβούν αρνητικές. Αλλά οι επαληθεύσεις δεν γίνονται στο τέλος, αλλιώς ε, προφανώς δικαίως διαμαρτύρονται οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Αντωνότσι. Ο κύριος Δελάντη. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών και εσάς κυρία Πρόεδρε, διότι επιταχύνατε τη διαδικασία της συζήτησης η οποία εν μέρει μας φέρνει και σε δύσκολη θέση, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως ε, με τη συνάδελφο Άουκεν, βρισκόμαστε ε, να συζητάμε συνέχεια το θέμα των αποβλήτων στο Λάτιο, λες και πρόκειται για μοναδική προτεραιότητα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε στην Ευρώπη. Πάντως ε, πρόκειται για κατεπίγουσα κατάσταση η οποία είναι συνεχής και ε, απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες και υπενθυμίστηκε και η περιοχή του Κορκόλε και την οποία είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες και ουσιαστικά έχουμε και πάλι το ίδιο σενάριο. Αυτό που μας είπαν οι εκπρόσωποι των πολιτών και οι συνάδελφοι προηγουμένως είναι ότι δημιουργείται μια θεσμική κακοφωνία που για έναν Ιταλό Ευρωβουλευτή που βρίσκεται εδώ είναι σχεδόν ε, όνειδος, διότι έχουμε μία σειρά από επίσημες αρχές οι οποίες είναι κατά της διαδικασίας, έχουμε μία σειρά από αρχές που πότε είναι υπέρ, πότε υπαναχωρούν, πότε επανέρχονται στην αρχική τους θέση ε, και ουσιαστικά γίνεται ένα παιχνίδι στο τέλος ε, αυτή που χάνει σίγουρα είναι η διαφάνεια και η... υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, την επιστολή του αρμόδιου επιτρόπου τη βλέπουμε με πολύ μεγάλη ε, ανησυχία ε, και για τη στάση που τήρησε ο επίτροπος ο Σιάνο, αλλά και γιατί δεν λέγεται και όχι τόσο σε εμά τους ευρωβουλευτές αλλά στους ε, ε, πολίτες της περιοχής του Ριάνο τους λένε ότι το Ριάνο ε, δεν είναι πλέον μεταξύ των εναλλακτικών εκδοχών και επομένω ή θα του το πούν οριστικά ότι έχει αφαιρεθεί από το πρόγραμμα ή θα πρέπει ε, αυτός ο επίτροπο ο οποίο δεν ήρθε παρόλο που τον είχαμε προσκαλέσει εδώ το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο να μην μπορεί να λέει ότι ε, όπως και να έχει εντάξει θα βγάλουμε το Ριάνο και θα σκεφτούμε κάτι άλλο. Είναι σαν να προσπαθεί να αποφύγει να επισέλθει στην ουσία τη σημερινή συζήτηση. Δημιουργείται λοιπόν μια θεσμική κακοφωνία η οποία χαρακτηρίζει το όλο ζήτημα ζήτημα των αποβλήτων. Τώρα, για την περιοχή του Κορκόλε, πριν από δύο μήνες ε, έγινε ψηφοφορία στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, στην οποία λέγεται ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2020 και μετά δεν θα πρέπει να υπάρχουν χιτά. Προτείνεται λοιπόν στο 2012 μία λύση η οποία ε, ξεφεύγει από όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δικαίω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προχωρά με τι πρωτοβουλίε τη, ξεκινά διαδικασίε επί παραβάση για το τι γίνεται με τη διαχείριση τη περιοχή τη ε, Μαλαγκρότα και εμεί στην περιοχή του Λάτιο ε, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε δρόμου που βάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον όχι μόνο περιττή, αλλά δεν θα έπρεπε καν να γίνονται τέτοιε συζητήσει βάσει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αν όντω δεν βρεθεί μια λύση, ο εκβιασμός είναι ότι θα βρεθούμε πνιχμένοι στα σκουπίδια και με αυτή την ε, διαστραμμένη λογική των σκουπιδιών ουσιαστικά αποφεύγουμε την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αποβλάτων το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε. Εμείς εδώ σε αυτή την ε, ε, αίθουσα τον Ιούνιο είχαμε ξεκινήσει μία συνάντηση με ένα Δήμο ο οποίος κατά 95% κάνει διαφοροποιημένη ε, συλλογή αποβλήτων, ε, υπάρχουν στις περιοχές διάφορα μοντέλα αριστείας. Υπάρχει λοιπόν μια λύση για το τι μπορούμε να κάνουμε. Επομένως εδώ μάλλον πρόκειται και για οικονομικά συμφέροντα διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία δυστυχώς είναι πολύ πιο ισχυρά από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και φυσικά και της λογικής. Να προσθέσω και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο αναφέρθηκε εν μέρη. Εγώ στην περίπτωση του Κορκόλε, είχα αναφέρει ότι θα έπρεπε ίσως να μάθουμε και τι γίνεται με την ιδιοκτησία της περιοχής. Εκεί είχαμε μία ανιώνυμη εταιρεία ελβετικού δικαίου ε, και οι ιδιοκτήτες ήταν αυτοί που θα έπρεπε να, να φτιάξουν το χώρο της υγειονομικής ταφής. Και εδώ όμως έχουμε ε, έναν ιδιοκτήτη ο οποίος ε, κατά σύμπτωση είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης ε, του χιτά της Μαλαγκρότα και πριν από κάποιου μήνε είχαν ε, υπάρξει επικρίσεις επί του ζητήματο αυτού. Είναι κάτι βέβαια το οποίο είναι καθόλου νόμιμο, ίσω και διάφωνο, αλλά σίγουρα είναι αρκετά περίεργο, είναι μια ανομαλία. Είναι σαν να λέμε ότι θα σου κλείσω αυτό, μην ανησυχεί, θα σου ανοίξω καινούριο. Και φυσικά όλο αυτό πόρα απέχει από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές όπως και τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τη συζήτηση τώρα του Καρκόλε, είχαμε και την παρουσίαση της ε, Επιτροπής ε, Κομαφίας ε, από την Ιταλική Βουλή που μας παρουσίασε ανησυχητικά στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή. Ο Υπουργό ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τα όσα παρουσιάστηκαν στη σχετική έκθεση και εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα η έκθεση αυτή να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Επιτροπής ε, για το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα, διότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να συζητήσουμε πιο διεξοδικά αυτή τη στιγμή, αλλά που σίγουρα αξίζει τον κόπο να συμπεριλάβουμε στην τεκμηρίωση ε, βάση της οποίας από εκεί και πέρα η Επιτροπή ε, θα αποφασίσει. Ένα τελευταίο στοιχείο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες, δεν είναι ρητορικό, ε, προσπαθούμε να κινηθούμε ενάντια σε πολύ ισχυρά συμφέροντα, σε ένα κόσμο μέσων ενημέρωσης που δεν μας βοηθάει και πάντα ε, η ενεργός ε, συμμετοχή ε, των πολιτών. Ελπίζω να μπορέσει σε αυτή την περίπτωση, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να αποτελέσει ισχυρό μας σύμμαχο και να βρούμε έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε δημόσια ζητήματα και κυρίως το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή μας. Ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους πολίτες οι οποίοι έθεσαν στην προσοχή μας ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αλλά και σεβάστηκαν με πολύ συγκεκριμένο και υπεύθυνο τρόπο τους χρόνους μας. Μας έδωσαν περαιτέρω πολύτιμα στοιχεία για εξέταση εκτός από αυτά τα οποία είχαν καταθέσει με, τον έγγραφ, με τα έγγραφά τους. Τα αιτήματά τους διατυπώθησαν εκ νέου και από τις παρεμβάσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκληση υπάρχει ένα έμεσο αίτημα να μείνει ανοιχτή η αναφορά για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στην Ιταλία. Ζητήθηκε επίσης να συμπεριληφθεί η περιοχή αυτή στο πρόγραμμα επίσκεψης που θα κάνουμε στα τέλη Οκτωβρίου. Θα το προτείνω στους συντονιστές οι οποίοι αυτοί πλέον θα αποφασίσουν για το τελικό πρόγραμμα αυτής της αποστολής. Υπάρχει επίσης ένα αίτημα βοήθειας θα έλεγα και από την αρμόδια Επιτροπή επί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, προς την οποία θα μεταφέρουμε εμείς όλα αυτά τα έγγραφα έτσι ώστε να υπάρξει μια γνωμοδότηση. Προσθέτω ότι και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και με το σύνολο του Κοινοβουλίου ξέρετε ότι το θέμα των αποβλήτων όχι μόνο στην Ιταλία αλλά σε όλη την Ευρώπη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες συνεργασίες που θα επιτρέψουν στην πρόταση λύσεων οι οποίες θα επιτρέψουν να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή από πλευράς ορισμένων χωρών των συγκεκριμένων οδηγιών και ρυθμίσεων. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει και τη διαδικασία επί παραλήψη. Ξέρετε ότι εδώ και χρόνια παρακολουθούμε την περίπτωση της Μαλαγκρότα στο Λάτιο. Υπάρχει επίσης και ένα αίτημα διευκρινήσεων που έχει κατατεθεί σχετικά με τον σεβασμό των διαδικασιών που ακολουθούνται για την, για την αξιολόγηση την περιβαλλοντική, κάτι το οποίο έχουν ζητήσει και οι πολίτες της περιοχής. Εμείς λοιπόν θα προσθέσουμε το τελευταίο μας αίτημα προς τις τοπικές αρχές να υπάρξει η δυνατότητα και άμεσης αντιπαράθεσης και επιβεβαίωση συνεπώς των παραβιάσεων των νομικών ρυθμίσεων στις οποίες αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια των παρεμβάνσεών σας. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη και από πλευρά του Κοινοβουλίου να ζητηθεί μια απάντηση σε αυτό. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι τελικά θα έχουμε την δυνατότητα με να πιέσουμε τις τοπικές αρχές, τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα κληθούν να πάρουν τις αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν έχουμε εκτελεστικές αρμοδιότητες, αλλά ως προς αυτές θα πρέπει να στραφούμε και να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά και θα συνεχίσουμε σύμφωνα με τα στάδια τα οποία προβια... Ε, σας παρουσιάσει. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Περνάω στο, στο επόμενο θέμα. Θέλετε το λόγο? Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και εκτός από το να έρθετε σε επαφή και με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και να ζητήσετε και την καταμέτρηση των ζημιών τις οποίες έχουμε υποστεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα την 1345-2009 και 46-2010 στο σημείο 16. Πρόκειται για αναφορές οι οποίες έχουν κατατεθεί από πλευράς δύο Πολωνών υπηκόων. Η μία είναι η Ρένα Ρογκώστα, πρόεδρος της Ένωσης Stop Odgrifce, για να σταματήσει η υπαίθρια εξόριξη, επιφανειακή εξόριξη άνθρακα, λιγνίτη μάλλον, στη Νότια Σιλεσία. Και έχουμε επίσης και εκπροσώπους των πόλεων Ρούμπιν και Γκούμπιν. Eh, do la parola Κρουσελόσκα. Έχουμε επίση και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρουτσέλοσκ. Ευχαριστώ κυρία ε, ε, Πρόεδρε. Είμαι η, η ε, δήμαρχος μία από τις ε, πόλεις οι οποίες εμπλέκονται. Είχαμε παρουσιάσει και πέρυσι αυτή την περίπτωση διότι ουσιαστικά διαπιστώσαμε ότι ατυχώς ε, δεν δόθηκε συνέχεια στα αποτελέσματα της υποθέσεως αυτής. Το 2009 οι ε, πολίτες είχαν καταψηφίσει κατά 90% ότι ε, η ερώτηση αυτή ήταν η πιο σημαντική α, ε, πρόβλημα ε, ψηφοφορία στην περιοχή μας και σε άλλες κοινότητες ε, υπήρξε αρνητική ε, ε, απόφαση αλλά παραβλέφθηκε και αγνοήθηκε τελείως. Έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει συζήτηση και υπάρχει μία, ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία επιφανείας και πρόκειται για πράξεις που αναλαμβάνονται από το, κυβόρνη, από την κυβέρνηση πέρυσι και ε, στα πλαίσια ενός προγράμματος μέχρι το 2030. Ε, έχει υιοθετηθεί στο Κοινοβούλιο το κείμενο αυτό που θα έπρεπε να προστατεύει ε, την κοινότητά μας. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν έχει βοηθήσει η παρέμβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των πολιτών. Γι' αυτό και υποβάλαμε αυτά τα έγγραφα διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να να προστατεύσουμε και τα αποθέματα ε, και η εξόριξη αυτών των αποθεμάτων λιγνίτη θα οδηγήσει σε μία καταστροφή των εμπλεκομένων περιοχών και όπως ξέρετε πολλά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή η εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι εις βάρος ε, των ε, κατοίκων, των κοινωνικών εταίρων και ουσιαστικά λαμβάνει μόνο χώρα γιατί έχουμε ε, ένα πολύ ισχυρό λόμπι υπέρ της χρήσεως άνθρακος στην Πολωνία. Πέρυσι οι ευρωβουλευτέ είχαν ζητήσει επισήμως διεπιστολής ε, από τον ε, πρόεδρο της Πολωνίας ε, να εκφραστεί η κυρία Γκέριγκερ, κυρία Πολάσκα και άλλοι πολλοί και όλοι οι Πολωνοί ευρωβουλευτές χωρίς όμως να λάβουν απάντηση και αυτό είναι περίεργο. Θεωρούμε ε, ότι στη συνέχεια ένα καλό σημείο ήταν ότι οι Γερμανοί ευρωβουλευτές καθώς και άλλοι ε, συναντήθηκαν με έναν Πολωνό Υπουργό και υποθέσαμε ότι θα μπορούσαν ξεκινήσει κάποια συζήτηση του θέματος ελπίζοντας ότι θα υπήρχε επανέναρξη του διαλόγου αυτού χωρίς όμως να δοθεί καμία συνέχιση στον διάλογο, συνέχεια στο διάλογο αυτό και γι' αυτό αποφασίσαμε να υπάρξει μία πανεθνική ε, σύσκεψη ε, για να ε, μπορέσουμε να κατακρίνουμε αυτή την εξόριξη επιφανίας του λιγνίτη ε, και να ακουστεί η γνώμη μας διότι ε, δεν θέλουμε να εξορίσετε ε, λιγνίτη στην περιοχή. Δυστυχώς όμως η έκφραση του εγχειρήματο δεν πήγε καλά. Ο πρόεδρος Ντόναλτ Τούσκ που τότε προωθούσε ένα άλλο ενεργειακό πρόγραμμα είπε ότι η Πολωνία προσπαθεί στην Ευρώπη Ευρώπη να προωθήσει ότι ο λιγνίτης που είναι πολύ πολύτιμο αγαθό ενεργειακό θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ενώ σε μια περίοδο όπου υπήρχε αρνητικό κρίμα για την πυρηνική παραγωγή ενεργείας καταψηφίσαμε μια εναλλακτική λίστη. Κυρία Πρόεδρε και κύριοι, όπως βλέπετε η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν μας μιλάει καν. Ακόμη και η ε, επιστολή η οποία εστάλει έμεινε αναπάντητη, γι' αυτό και επανήλθαμε. Και παρουσιάσαμε αυτό, αυτή την ε, αναφορά διότι ε, θα σας προσκαλούσαμε να ε, επισκεφτείτε την Πολωνία να καθορίσετε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαν να υποβληθούν στην κυβέρνηση για να ξεκινήσει βάσει αυτών η κυβέρνηση μία συζήτηση με τους πολίτες πράγμα το οποίο θα ήταν πολύ θετικό και θα δώσω τώρα το λόγο στο συνάδελφό μου που είναι δήμαρχος της περιοχής Γκούμπιν. Τώρα δίνω το λόγο στον δήμαρχο αυτής της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, δεν είμαι μόνο εκπρόσωπος της ε, επαρχίας Γκούμπιλ αλλά συγχρόνως ε, ε, και πρόεδρος της ομάδος για το, ο, τις συμμαχίες για του συνασπισμού για το περιβάλλον στην Πολωνία και εδώ αναφερόμαστε ε, για την κοινότητα του Γκρόμπι και την περιοχή του Γουμπούσκι όπου το 2009 οργανώθηκε ένα δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα όμως του δημοψηφίσματος αυτού δεν ελήφθη υπόψη από την κυβέρνηση και στην περίπτωσή μας το Μάρτιο του 2012 ένα, υιοθετήθηκε ένα ε, περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει την προώθηση ε, της ε, εξορίξεως του λιγνίτη σε ορυχία επιφανείας χωρίς να υπάρχει ένα πρόγραμμα ή κάποια περιβαλλοντολογική μελέτη επιπτώσεων και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι άποψεις οι απόψεις των πολιτών. Στη Γερμανία υπάρχουν ε, ήδη ε, δύο ε, στραθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας που χρησιμοποιούν άνθρακα και στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη δύο οι οποίοι εκπέμπουν πολύ υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακο στην ατμόσφαιρα. Εάν λοιπόν προσθεθεί σε αυτούς άλλος ένας θα υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ε, διοξιδίου του άνθρακος εάν τρεις, ε, τρεις ε, σταθμοί και είναι άνθρακα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να σκεφτούμε τι θα γίνει στο περιβάλλον. Θέλουμε να τονίσουμε επί του προκειμένου ότι έχουμε έξι περιοχές σε αυτή την περιοχή που προστατεύονται από τη Natura 2000 σε μεγάλη έκθεση και αυτή η ε, έκβαση θα ε, ε, επηρέαζε αρνητικά τις περιοχές αυτές και πέραν αυτού υπάρχουν και διάφοροι ε, οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι μας πιέζουν να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα για να εξασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό και είναι βασικό η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, εξηγήσει πόσο σημαντική και δύσκολη είναι η κατάσταση διότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και άλλες περιοχές στην ε, χώρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι Τόμας Βεσνιεύσκη, ε, Προσωπώ την Επιτροπή ε, σταματήστε τη ορυχεία επιφανίες και συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν. Έχουμε διαμαρτυρηθεί ε, κατά της, ε, του γεγονότος ότι αγνοήθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και αυτό έχει ε, σχέση και με την προστασία ε, της βιομηχανίας ή στην Πολωνία αλλά προσπαθούμε συγχρόνως να προστατεύσουμε και τον ενεργειακό τομέα όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και μπορούμε και δεν είναι δυνατόν να βασιζόμαστε σε ε, κάψιμα όπως ο λιγνίτης και ο άνθρακας που προκαλούν μεγάλη ρήπανση και ε, μετατοπίζουν και μεγάλες ε, ομάδες πληθυσμών και υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι κινούνται αντίθετα σε συμφέροντα πολλών πολιτών εξού και ε, ε, προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέραν των ενεργειών ή στην Πολωνία πέρυσι ε, τον Ιούνιο είχαμε κάνει δύο διασκέψεις προωθώντας την, ε, την εξόριξη ε, του, του, λιγνίτη αλλά όχι σε ορυχεία επιφανίες που είναι μία πεπαλαιωμένη μέθοδος και απευθυνθήκαμε στις αρχές οι οποίες όμως ε, με μεγάλη υπεροψία μας αγνόησαν. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξετε ε, το θέμα αυτό, να το μελετήσετε και παρακαλούμε να δεχθείτε την πρόσκλησή μας. Ελάτε στην Πολωνία να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπρέκλαντ, εξ ονόματος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, συζητήσαμε την αναφορά αυτή πέρσι στις 15 Ιουνίου, από περιβαλλοντική σκοπιάς ε, θεωρήσαμε ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Μία διαδικασία βάσει της οποίας ε, θα γινόταν στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ενεργειακή πολιτική της Πολωνίας μέχρι το 2030 και όπως σας είχα εξηγήσει και πέρσι δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης της σχετικής οδηγίας. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιες επικρίσεις για το γεγονός ότι η ημερομηνία διαβούλευσης ε, στην ιστοσελίδα δεν ήταν σαφής, αλλά οι δήμαρχοι μπόρεσαν να διαβιβάσουν τις απόψεις τους και ε, απόδειξη αυτού είναι ότι υπήρχε και το αρνητικό δημοψήφισμα με ποσοστό πάνω από 90%. Ε, και από εκεί και πέρα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορεί να υπάρχει παραβίαση της οδηγίας για του φυσικού οικοτόπου και μπορεί να καταστρέφονται βάσει αυτής της διαδικασίας ε, χώροι του Natura 2000. Πέρσι σας είχα πει ότι είχαμε κάποιες ενδείξεις από τις πολωνικές αρχές ότι επ' αυτού υπήρχε σαφής δέσμευση να μην γίνουν επενδύσεις ε, ε, σε νέα ορυχεία μέχρι το 2030 και κατόπιν ετήματός σας ζητήσαμε και επιβεβαίωση από τις πολωνικές ε, αρχές ε, για αυτές τις μηδενικές επενδύσεις και αντίθετα από τα όσα μας λέτε εσείς πήραμε την επιβεβαίωση από τις πολωνικές αρχές υπάρχει επιστολή με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2011 με υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος που λέει ότι δεν θα υπάρξουν εξοριστικές δραστηριότητες στην περιοχή μέχρι το 2030. Από δική μας λοιπόν περιβαλλοντική σκοπιά, το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν εξορυκτικές δραστηριότητες είναι θετικό στοιχείο. Θα θυμάστε ίσως ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια περίπτωση που αφορούσε την ε, Ελλάδα ε, στην 2 ε, κάθετος 10 ε, απεφάνθη ότι μπορεί κάλλιστα κάποιο να σταματήσει όλε τι δραστηριότητε σε ένα χώρο που προστατεύεται από το Natura 2000 ε, και επομένω εμεί θεωρούμε ότι έχουμε λάβει αυτό που επιθυμούσαμε εφόσον δεν θα υπάρχει καμία εξορρεκτική δραστηριότητα. Από ό,τι κατάλαβα έχει παγώσει οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή. Ε, και όλες οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες θα μπορεί με να ανασταλούν, αλλά αυτό που μας ενδιέφερε από πλευράς περιβάλλοντος ήταν να προστατεύσουμε ε, χώρους προστατευόμενους από το Natura 2000 και βάσει της επιστολής ε, της πολωνικής κυβέρνησης, την οποία μόλις σας ανακοίνωσα, διότι εσείς δεν πήρατε απάντηση στη δική σας την επιστολή, από περιβαλλοντική σκοπιά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντάξει. Όπω σα είπα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από του Δημάρχου. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το λύσουμε εμεί μέσω περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά υπάρχει ίσω η δυνατότητα επίσκεψης της Επιτροπής σας επιτόπου και ίσω αυτό να επαφίεται σε εσά, να είστε εσεί οι οποίοι θα διαβιβάσετε το μήνυμα τη δικαιοσύνη και τη χρηστή διακυβέρνηση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και η συνεργασία μεταξύ δημάρχων και κεντρική κυβέρνηση. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέριγκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα συμφωνήσω με τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τα πράγματα. Αν δει κανεί τον κοινοτικό νόμο, θα δει ότι ό,τι έγινε μέχρι τώρα είναι σύνομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υπογραμμίσει ότι απαιτείται για τέτοιου είδους επενδύσεις ε, ε, ενημέρωση, διαβούλευση και τι καλύτερη καλή διαβούλευση μπορεί να φανταστεί κανείς από ένα δημοψήφισμα όπου το σύνολο των κατοίκων της περιοχής αποφασίζει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να προχωρήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ορυχεία στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πολλά χρήματα των διαθροτικών ταμείων έχουν επενδυθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και στόχος μας θα πρέπει να είναι να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των επενδύσεων αυτών και γιατί σταθερότητα μπορούμε να μιλάμε αν ξαφνικά οι επενδυτές αποχωρούν και ποιος θα αποφασίσει να επενδύσει σε μια περιοχή όταν η περιοχή αυτή από τη μία μέρα στην άλλη καθίσταται απαρχαιωμένη. Ε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λοιπόν την πρόταση για, για το δημοψήφισμα και όταν δει κανεί την κοινοτική νομοθεσία αλλά και σε πολλές χώρες υπάρχει η μέθοδος ε, η δημοψηφισματική και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραβίαση του νόμου ε, επέρχεται όταν ε, η δίκαιη έκφραση της λαϊκής βούλησης αγνοείται. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα από τους αναφερομένους ένα πράγμα, αν θα μπορούσαν να κάνουν κάποια επιπλέον σχόλια και να μας πούνε αν γνωρίζουν ότι έχουν υπάρξει στην Πολωνία και άλλα δημοψηφίσματα τα οποία αγνοήθηκαν και αυτά Πρόκειται για μια τακτική θα έλεγα πρακτική. Τι είναι αυτό το οποίο ε, επηρεάζει τις εξελίξεις στην περιοχή αυτή. Έχουν υπάρξει άλλες επενδύσεις με ευρωπαϊκά χρήματα. Ε, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην τιμή των γεών και της κατοικίας. Υπάρχουν μεταναστευτικά ρεύματα εκτός περιοχής. Ποιες είναι οι συνέπειες γενικά γιατί θα ήθελα να πω ότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα αυτό, κάποιες διαδικασίες έχουν παγώσει και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της περιοχής και στις μελλοντικέ της εξελίξεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν οι αναφερόμενοι μπορούν να μας δώσουν κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Κυρία Κολάρσκα, έχεις δει στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ένα πρόγραμμα ε, επισκέψεως στην Πολωνία και κατά αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε αμφιβολία θα μπορούσε ε, να διασκεδαστεί διότι νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα και να δούμε και την ανάπτυξη της περιοχής και τον προγραμματισμό της ε, επαρχίας και της εθνικής κυβέρνησης. Για ας το περιλάβουμε λοιπόν στο πρόγραμμά μας. εντωμεταξύ. όμως είπατε ότι είναι βρώμικη ενέργεια, ότι θα ρηπαίνει, θα υπάρξει ρήπανση στην περιοχή σας. Έχετε αναπτύξει κάποια άλλη πηγή ενεργείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν μία ερώτηση και μία ανακοίνωση. Στην Επιτροπή μας είμαστε όλο και πιο πιεσμένοι από το πρόβλημα των, ε, της ελλείψεως ενεργειακών πόρων, γι' αυτό και ανοίγουν όλο και περισσότερα ορυχεία και ε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες στον τομέα αυτό και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, αλλά δεν πρέπει μια τέτοια ενέργεια να είναι εις βάρος του περιβάλλοντος. Μία, ένα ορυχείο επιφανείας πολλές φορές είναι μια ενα ορυχειο επιφανιας πολλες φορες καταστροφή. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για, τις, ε, για να περιοριστούν οι, ε, οι οικολογικές ε, ζημίες. Μπορεί να υπάρξει άλλου τύπου εξόριξη και όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής αυτής εξαρτάται από αυτό το ρηχείο υπάρχουν άλλες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης χωρίς να χρησιμοποιηθεί αυτό το ορυχείο. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι έχω μία ομάδα Ολλανδών οι οποίοι παρίστανται στις εργασίες της ε, Επιτροπής μας ε, για να παρακολουθήσουν πώς ε, λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Ε, θα ε, εποφεληθώ ότι μπορώ να μιλήσω δανέζικα και καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστώ γιατί ε, συζητείτε αυτό το θέμα διότι όπως ήδη ελέγχθη δεν είναι ε, αποδεκτός ο τρόπος αυτός εξορίξεως. Υπάρχει μία υπεροψία έναντι της φύσεως, έναντι του τοπίου, του περιβάλλοντος ε, και ε, αυτή η μορφή εξορίξεως θα έπρεπε να καταργηθεί. Αλλά πολλές φορές ε, λέει η Πολωνία ότι δεν θέλει να προσαρμοστεί ε, σε νέες τεχνολογίες, δεν θέλουν να προωθήσουν πιο βιώσιμες ε, πηγές ενέργειας, θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες επιδοτήσεις για πεπαλαιωμένες μορφές εξορίξεως ενεργειακών πηγών και θα έπρεπε να αλλάξει και η νοτροπία της βιομηχανίας σχετικά με την προμήθεια ενεργείας στην χώρα αυτή. Δηλαδή η Πολωνία μόνη της θα χρειαστεί να αποφασίσει πότε θέλει να προσχωρήσει στις σύγχρονες χώρες και πότε θέλει ε, να ε, τραβήξει μια γραμμή για τις ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον. Όλα αυτά μπορούμε να τα σημειώσουμε, αλλά εγώ αφισβητώ αν όντως μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει μία σωστή μελέτη περιβαλλοντολογικής αξιολογήσεως. Δηλαδή νομίζω ότι ούτε οι ε, πολίτες δεν θα το γνωρίζουν. Θα έγινε κάτι ε, και κλεισμένο το θυρών και θα φτάσει το 2013, θα χρειαστεί ε, αυτό το θέμα να εφαρμοστεί και μέχρι τότε η κάτοικοι της Πολωμίας έχουν ε, χρόνο να ε, προωθήσουν τα θέματα, να προσχωρήσουν στη σύγχρονη κοινωνία και να μην καθυστερούν τα πάντα, διότι η Πολωνία είναι μια χώρα η οποία ε, χρησιμοποιεί τη φτώχεια της σαν μια δικαιολογία για να μην εξυγχρονιστεί. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά η Πολωνία είναι γειτονική χώρα και προς τη Δανία και εγώ ευχαρίστως να σα στηρίξω εν ονόματι ε, της κυβέρνησης της Δανίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ε, αλλά όλα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Έχω και μία ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είσαστε ικανοποιημένοι με την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που έχουν γίνει και ενεπλάκησαν οι πολίτες σε αυτό το έργο. Η κυρία Κολάσκα ζητάει το λόγο. Ναι, εγώ γνωρίζω απόλυτα το θέμα αυτό και με τον συνάδελφο Πιότρ Μπόρις ε, το έχω συζητήσει επανειλημμένως διότι προέρχεται από την περιοχή. Δεν έχει ληφθεί απόφαση και εμείς διαμαρτυρόμαστε κατά της απόφασης. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι είναι όλα θολά. Το θέμα αυτή τη στιγμή εκκρεμεί δεν διαμαρτυρόμαστε εμείς για ηλυμένη απόφαση. Υπάρχει σειρά από ε, σχέδια τα οποία εκκρεμούν και αυτό είναι αυτό το οποίο πάμε να επιβεβαιώσουμε στην αποστολή μας ε, στην Πολωνία. Ε, εγώ δεν λέω ότι αυτό το καθεστώς είναι θετικό, ίσα ίσα λέω το αντίθετο, ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφήνεια είναι εις βάρος της περιοχής. Η ναι, η απόφαση να σταματήσει η εξόριξη ε, λιγνίτη έχει, είναι λιμένη. Δεν θα υπάρξει ε, καμία νέα υποδομή ε, άνθρακα, αλλά θα υπάρξουν άλλα λιγνητορυχεία. Η συνάδελφο μου ζήτησε να μιλήσω για τι νέε τεχνολογίε. αν οι ήπιες μορφέ ενέργεια μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή εκείνη. Ναι, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά δεν λαμβάνονται άδειε ε, για να ε, προχωρήσουν τα σχέδια, γιατί τα πάντα πρέπει να γίνονται με βάση τον άνθρακα. Και γιατί αυτό, διότι υπάρχουν ισχυρέ ομάδε πίεση, οι οποίε πιέζουν τι τοπικέ αρχέ. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θα διευκρινίσουμε στην ε, επίσκεψη που θα κάνουμε στα τέλη Οκτωβρίου. Πρέπει να δούμε τα πράγματα η διεισόμαση διότι πρόκειται για ε, στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με λόγια. Ίσως ε, να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερο και από τους αναφέροντες. Ε, η πρόεδρος να δώσει το λόγο στους αναφέροντες για να απαντήσουν, χωρίς μικρόφωνο αναφέρει. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν. Ένα αφορά τα υπόλοιπα δημοψηφίσματα τα οποία έγιναν στην Πολωνία. Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, σε μια μικρή ε, πόλη στη Βόρεια Πολωνία, στον Κόνσκι, έγινε ένα δημοψήφισμα για ε, το άνοιγμα πυρηνικού εργοστασίου στην ε, Πολωνία, στην περιοχή. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έγινε απόλυτα σεβαστό. Το έλαβε υπόψη του και ο Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ακούσουμε την κοινή γνώμη και ο λόγος των πολιτών ε, ε, αξίζει ε, όσο τίποτα άλλο, αλλά ποτέ δεν ακούσαμε κάτι αντίστοιχο για το δικό μας το δημοψήφισμα. Εμείς ε, δεν λάβαμε ποτέ διάψευση για το πρόγραμμα της κυβέρνηση να ανοίξει ε, αυτό το ορυχείο, το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι ε, τα ορυχεία αυτά λιγνίτη και άλλες περιοχές ε, θα περιληφθούν σε ένα πρόγραμμα υποδομών το οποίο δεν σχετίζεται απαραίτητα με τον τομέα της ενέργειας. Κατόπιν είχαμε και μία ερώτηση για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Στην περιοχή του Γκούβιν, από την οποία προέρχομαι, στην ε, επαρχία του Λουμπούσκε, προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις ε, στην εξόριξη λιγνίτη. Και εδώ και ένα χρόνο υπάρχει ανοιχτή διαμάχη με τις τοπικές αρχές, ε, υπάρχει μια περιοχή ε, στο Δήμο μας και υπάρχει και επενδυτές ο οποίος κατόρθωσε να πείσει τις τοπικές αρχές ότι ο μόνος δρόμος είναι ο Λιγνίτης και ακόμα βρισκόμαστε λοιπόν σε αδίέξοδο. Όσον αφορά λοιπόν ε, το δικό μου το Δήμο τώρα, λέω τρίτος αναφέρον, εκκρεμούν ακόμα 44 αποφάσεις ε, που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία ε, ιδίου αριθμού πυρηνικών σταθμών. Οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα διότι δεν μπορούν να προωθήσουν ε, σχέδια εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Όσον αφορά τώρα... Υπάρχουν ε, πρόβλημα με τις τουρμπίνες ε, οι οποίες επειδή κυκλοφορούν εκτορύβες στην περιοχή παγιδεύονται και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Ε, εσύ Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Νομίζω ότι προ το παρόν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Η απόφασή μα είναι να παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα, διότι εκκρεμεί φυσικά όλο. Ευτυχώ μία από τι δύο περιπτώσει δεν είναι επίγουσα, επομένω μπορούμε Εάν οι συνάδελφοι συμφωνούν, μπορούμε να αναστείλουμε οποιαδήποτε απόφαση η οποία θα ληφθεί μετά από την επίσκεψή μα, διότι είναι ήδη προγραμματισμένη η διερευνητική επίσκεψη επιτόπου ε, στις περιοχές ε, που ε, αναφέρονται στις ε, αναφορές και θα γίνει αξιολόγηση από εκεί και πέρα στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει μετά από την επίσκεψή μας. Δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση στο σημείο αυτό και ε, αναβάλουμε την απόφασή μας ε, για ε, μετά από την επίσκεψή μας. Ευχαριστώ τους αναφέροντες και να περάσω στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την αναφορά της κυρίας Μαρία Λουίζα Ριβέρα Άλβαρεθ, Ισπανικής Ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ασοσιαθιών Δεβεθίνος Βαλντορέμπλο στο Αρνάδο της Λεόν. και ε, το αντικείμενο της αναφοράς είναι οι καταστροφικές επιπτώσεις ε, των ορυχείων επιφανείας ε, σχιστόλιθο που λειτουργούν παράνομα στο χωριό Αρνάδο. Δεν είναι παρούσα η αναφέρουσα, επομένως να δώσω απευθεία το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ράμος Φλωρίδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το αντικείμενο αυτής της αναφοράς είναι μία σειρά το αντικείμενο της αναφοράς είναι μια σειρά ε, ορυχεία σχιστόλουθου στην περιοχή της Καστίγια Ελαιών ε, στην ε, Ισπανία. Η αναφέρουσα καταγγέλει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και για τις πιθανές ε, επιπτώσεις στην ασφάλεια των ατόμων των συγκεκριμένων ορυχείων. Να ε, σας πω ότι πρόκειται για παράνομα λατομία και προβλέπεται και επέκτασή τους και καταγγέλλεται και το γεγονός ότι οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές ε, αδρανούν. Ε, έγινε και καταγγελία στον εισαγγελέα της ε, αυτόνομης περιοχής της Καστίγια Λεών και ε, πρέπει να πούμε εδώ ότι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μελέτησαν την αναφορά την οποία διαβίβασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα με βάση το κοινοτικό δίκαιο σε θέματα περιβάλλοντος, ε, διότι πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο αφενός υπάρχει περιβαλλοντική κοινοτική νομοθεσία η οποία ε, εφαρμόζεται, αλλά υπάρχουν και θέματα ε, εξόριξης και εκμετάλλευσης ορυχείων στην Ισπανία που δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι η σχετική οδηγία για την ε, ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη γνωστή 97 85337, η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 9711. Και εδώ έχουμε εφαρμογή του παραρτήματο 2 τη οδηγία για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει που αναφέρεται στο σημείο 2α και αφορά τα ορυχεία και τα λατομεία στα προγράμματα ε, που περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση. Όπως ξέρετε, βάσει του παραρτήματος 2, τα όσα περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 δεν υπόκεινται πάντα σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως γίνεται με το παράρτημα 1 και εξαρτώνται και από τα κριτήρια τα οποία έχει εφαρμόσει η αρμόδια αρχή μεταφοράς της οδηγίας και την ε, περίπτωση όπως για παράδειγμα το μέγεθος, τις σχετικές επιπτώσεις κλπ. Ε, οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν και τι γίνεται με την κοινωτική νομοθεσία προστασία του περιβάλλοντο, ε, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για του φυσικού κοτόπους που εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχουν ε, αρνητικέ επιπτώσει στο δίκτυο Natura 2000 που δεν φαίνεται ότι υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από την εξέταση της αναφοράς και για να την αντιμετωπίσουμε καταλήλω, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία έρευνας, η οποία περιλαμβάνει, όπως σας είπα, μόνο το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Έγινε μια ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιε ισπανικές αρχές. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ζητήσει σε αρκετέ περιπτώσει πληροφορίε από τι αρμόδιε Ισπανικέ Αρχέ σχετικά με τα μέτρα τα οποία ενέκριναν προκειμένου να τηρήσουν την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πληροφορίες για το τι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση και για το συγκεκριμένο λατομείο σχιστόλιθου που αφορά του αναφέροντες. Για να συνοψίσω και να είμαι λίγο πιο λακωνικός, ε, λάβαμε απάντηση από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές. Ε, υπάρχουν εκθέσεις ε, από το Περιφερειακό Διαμέρισμα Περιβάλλοντος της Καστίγια Το τμήμα τουρισμού επίσης ε, έχουν αποσταλεί και από τα δύο από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Ορυχείων. Η συγκεκριμένη εκμετάλλευση, το συγκεκριμένο ορυχείο έχει άδεια ε, για 10 χρόνια και υπάρχει και ένα σχετικό πρόγραμμα αποκατάστασης ε, επειδή υπήρχαν βέβαια διαμαρτυρίες από τους περίοικους ε, οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έκαναν αρκετές επιθεωρήσεις κυρίως για τον έλεγχο της διαχείρισης των απορριμμάτων και τι γίνεται ε, με τα πυρήματα του λατομείου και ε, υπήρξαν μια σειρά από προϋποθέσεις και κυρώσεις ε, προς το συγκεκριμένο λατομείο. Το 2011 αποφασίστηκε να κλείσει τμήμα των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένη εκμετάλλευσης. Ξεκίνησαν διάφορες διαδικασίες κυρώσεων κατά της επιχείρησης, διότι δεν είχε τηρήσει πλήρως την άδεια όπως της είχε δοθεί και η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα να συνεχίσει την εξορεκτική της διαδικασία και από εκεί και πάει λάβει και σχετική παράταση της άδειας που έχει. Είναι ε, αυτή τη στιγμή ε, υποεξέταση μαζί με τη μελέτη περιβαλλοντικών υποστό, επιπτώσεων με βάση και την ομοθεσία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυτόνομης περιοχής. Ε, πρέπει επίσης να πω ότι ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής ασχολήθηκε με την υπόθεση και μετά από παρέμβασή του οι αρχές της αυτόνομη περιοχής δραστηριοποιήθηκαν λίγο περισσότερο και πήραν μια σειρά από μέτρα και έτσι ο Ευρωπεριφερειακός Διαμεσολαβητής ε, αρχιοθέτησε την υπόθεση και θεωρεί ότι έδρασαν σωστά οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας ε, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μια τελευταία απάντηση που λάβαμε από τις Ισπανικές Αρχές ε, με ημερομηνία Απριλίου του 2012 μας έλεγε ότι είναι εξελίξη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ορυχείου και φυσικά ότι υπάρχουν και μέτρα ε, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των περίοικων που ζουν ε, κοντά στην ε, συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Με βάση λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες και λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως σας είπα και προηγουμένως, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μόνο την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεν μπορέσαμε σε αυτή την περίπτωση να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει παραβίαση κοινοτικού δικαίου ε, σε θέματα περιβάλλοντος. Θεωρούμε όμως ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές λαμβάνουν μια σειρά από μέτρα ώστε να βεβαιωθούν ότι εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ κύριε Άουκερ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεν νιώθω ασφαλής από αυτά τα οποία άκουσα. Εγώ είδα ακριβώς αυτό το λατομείο στα βόρεια της Λεών εδώ και λίγα χρόνια κοντά στις Αστούριας και ήταν καταστροφικό στην ουσία. Έσκαβαν την κορυφή του βουνού. Και στην ουσία δεν ήταν χρησιμοποιήσιμο το συγκεκριμένο προϊόν Ξέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τέτοιου είδους ε, ορυχία στην Ισπανία, πάντως η διαχείριση της κατάστασης από τις τοπικές αρχές ήταν καταστροφική, για να μην πω τίποτα περισσότερο. Απαιτείται να το εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι η ενημέρωση την οποία έχουμε, και δεν κατηγορώ την Επιτροπή γι' αυτό, δεν είναι επαρκές. Ο αναφερόμενος θεωρεί ότι οι παράνομες δραστηριότητες συνεχίζονται. Μέιερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που μας έδωσε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εκρεμεί η διαδικασία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επομένως θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να δούμε αν όντως ε, αυτή η διαδικασία θα έχει θετική έκβαση και ότι το συγκεκριμένο ορυχείο τηρεί όλες τις ε, διατάξεις Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Καλώς νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν με τη συγκεκριμένη απόφαση να λάβουμε υπόψη μας την αναφορά αυτή για να περιμένουμε και την κατάληξη της διαδικασίας την οποία έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μείνουμε ενήμεροι για τις εξελίξεις. Περνώ λοιπόν τώρα στην επόμενη αναφορά 980 στο σημείο 18 από πλευράς του κυρίου Τόρκιλντ Τόντσεν, εξ ονόματος της ομάδας πολιτών Μποργεν γιατί για το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου ανάμεσα στο Κίπλευ και στο Σόντεβοργκ. Δεν είναι ο αναφέρον εδώ και γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο και για τη συγκεκριμένη αναφορά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η θέση της Επιτροπής ε, είναι η εξή. Στο παρελθόν υπήρχε μια δυνητική παράβαση από πλευράς Δανίας για τις διαδικασίες. Στείλαμε μια επιστολή επίσημη προειδοποιητική. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες των αρχών της Δανίας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, από τον αυτοκινητόδρομο που περνά κοντά στον τόπο αυτό που είναι Natura 2000. Ε, παίρνουν μέτρα για την προστασία των βατραχοειδών και ταυτόχρονα ο θόρυβος του νέου αυτοκινητοδρόμου επί των πτηνών είναι ελάχιστος. Δεν υπάρχει λοιπόν επίπτωση για το περιβάλλον. Για μας λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχουν παραβιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Hogan. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι αξιοπερίεργο ότι η Επιτροπή απαντά έτσι. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ε, σχετικά με τις επιπτώσεις διότι αυτό δεν έγινε στη Δανία, διαφοροποιήθηκε η αξιολόγηση και δεν εξετάσαμε τη συσσόρευση. Αν δούμε λοιπόν τον χάρτη βλέπουμε ότι αυτές οι περιοχές ε, είναι συνδεδεμένες και βλέπουμε ότι υπάρχει μία, ε, μία επιδείνωση λόγω και της ατμοσφαιρικής ρηπάνσεως. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε ολόκληρο το φάσμα και όχι να τοποθετούμαστε μόνο σε ένα σημείο το οποίο οποίο μπορεί να μην έχει επιπτώσει στην Natura 2000. Ε, πέραν αυτού πιστεύω ότι η δανική κυβέρνηση αρχέτος του χρώματός της ακόμη και αν η προηγούμενη ε, κυβέρνηση ε, όταν ερωτήθηκε είπε ότι όλα πήγαιναν καλά και ότι τέτοιοι δρόμοι έπρεπε να κατασκευάζονται δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει να μείνουμε με δεμένα χέρια στην ε, ε, Δανία και ε, ό,τι έγινε έγινε τώρα για τα μελλοντικά όμως προγράμματα θα έπρεπε να φροντίσουμε η οδηγία να, ε, ε, να γίνεται σεβαστή ζητά να εξετάσουμε όλες τις πτυχές για τις διόδους οι οποίες δημιουργούνται και για τα μέτρα η κατάσταση είναι εξίσου κακή όπως και στην αρχή όταν ζητήσαμε να κρατήσουμε κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Δεν ξέρω αν ε, κάτι μπορεί να γίνει επ' αυτού. Μπορούμε απλούστατα να πούμε ακόμη ότι είναι δυνατόν ε, να συμπεριφέρεται κανείς έτσι εις την έναντι των, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και υπάρχουν εξαιρετικές ε, οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται 100%. Η Δανία έχει πόρους ακόμη και αν ε, η κυβέρνηση πάντοτε παραπονείται ότι ε, είναι εποχή ρητότητος. Ε, εκπρόσωποι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν με ικανοποιεί διότι θεωρώ ότι δεχθήκατε ελαφρά την καρδία αυτές τις δικαιολογίες της Δανίας και δεν θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει. Ο υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει ότι έχει γίνει αξιολόγηση. Εάν όμως η κυρία Άουκεν ε, έχει, έχει κάποια αντίρρηση. Εμείς έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στον Δανό Υπουργό Περιβάλλοντας, αλλά αν θέλετε να τον ξαναρωτήσουμε. Πιστεύω ότι βάσει αυτών των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, των σχολείων της κυρίας Όκεν δεν υπάρχουν πλέον άλλες παρεμβάσεις και μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά και εν πάση περιπτώσει να ζητήσουμε όχι με συγχωρείτε, χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι μπορεί να υπάρξει μία νέα αίτηση. Ε, ε, τι έχει γίνει διότι δεν νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι ε, και θα μπορούσαμε να το κλείσουμε γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε γενικά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Μπορούμε να διατηρήσουμε ανοιχτή ε, την αναφορά και να μείνουμε μία άλλη πιο ε, επακριβή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάξει, ωραία. Ωραία, οπότε διατηρούμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η αναφορά υπαριθμών 0323 ε, του 2011 του κυρίου Αλεχάνδρο Σάντσες και για την αναφορά αυτή παρίσθεται ο κύριος Λόπες Ντεουράλ Δεγαρμεντία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν είναι δευτερεύον ζήτηση, ζήτημα. Ε, στοιχίζει χιλιάδες νεκρούς κάθε χρόνο, προβλήματα για την οικονομία μας και την υγεία μας και χρειάζονται μόνιμα μέτρα προκειμένου να μειωθεί. Πρόκειται για το Δήμο της Μαδρίτης πρόκειται για μία από τις περιοχές τις οποίες έχουμε την περισσότερη ατμοσφαιρική ρήπανση και επειδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία της ρήπανσης ε, στη Μαδρίτη από το 2011 και μετά, ε, ξεκίνησε μια διαδικασία καταγγελίας, λάβαμε κάποια στοιχεία, ε, είχαμε απάντηση και λέγεται ότι υπήρχε δυνατότητα να ε, μεταφερθούν οι σταθμοί μέτρησης ε, σε περιοχές κοντά σε πάρκα κλπ, ώστε να μπορέσει να δώσει πιο ευνοϊκά στοιχεία. Βέβαια, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε και οι 19 από τους 24 σταθμούς βρέθηκαν στην ε, να καταγράφουν στοιχεία περίπου στα όρια ε, διοξιδίου του αζότου και παρά το γεγονός, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλά ε, βρίσκονται κοντά σε πάρκα. Ο αριθμός των σταθμών που λειτουργούν περισσότερο αυξήθηκε από 6 έως 9. Η περιοχή η οποία πλήττεται περισσότερο είναι η κεντρική περιοχή της Μαδρίτης και το 2012 η κατάσταση συνεχίθηκε η ίδια. Στις ε, ε, πρώτες ενδείξεις ε, ελέγχθη ότι η Μαδρίτη τηρεί την ομοθεσία ε, υπήρξαν και κάποιες όμως μετρήσεις που έδειξαν ότι σε πάρα πολλούς μήνες ε, βρισκόμασταν πάνω από τα όρια ε, σε ορούμενα ή διαδιοξίδιο του αζότου και όζων παρά το γεγονός ότι επιτρέπονται ε, να υπερβούν τα όρια ελάχιστες φορές μέσα στο ένα έτος είχαμε και μήνες ολόκληρους. Από τα καταστρεπτικά στοιχεία ρήπανσης λοιπόν που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια η Μαδρίτη, η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν ε, τον αέρα της Μαδρίτης και πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο ε, κατά βάση ε, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται ε, είναι απλώς προληπτικά, λαμβάνονται κάποια μέτρα τα οποία σε κάποιες ώρες της διάρκεια της ημέρας προσπαθούμε να μειώσουμε τα όρια δεν ε, φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να περιορίσουν ε, τη ρήπανση, δεν περιορίζεται καθόλου η κίνηση στην πόλη, δεν υποστηρίζεται καθόλου η χρήση πολυδηλάτου, ούτε ε, η μείωση της κίνησης σε περιοχές όπου έχουμε υψηλά ποσοστά και αυτό το σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε ε, περιλαμβάνει μέτρα κατά την άποψή μας. Και επίσης υπάρχουν και μια σειρά από μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ε, διότι θεωρείται ότι η κυκλοφοριακή κίνηση είναι το βασικό στοιχείο ρήπανσης ε, και ε, παρόλα αυτά ο Δήμος της Μαδρίτης ε, θα σταματήσει τις ενισχύσεις της, ε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αύξηση ε, στη χρήση και ο καθένας θα χρησιμοποιεί περισσότερο το ιδιωτικό του αυτοκίνητο όχημα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τις οικογένειες αλλά και στη στρατηγική για τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρξουν μειώσει λοιπόν στο κόστος των υπηρεσιών των μέσων μαζικής μεταφοράς, ε, ενώ στην πραγματικότητα θα οδηγηθούμε σε αύξηση, διότι μέχρι τώρα υπήρχε επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς ε, και ε, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ρήπανση. Και όλα αυτά φυσικά οφείλεται ε, στα μεγάλα προβλήματα, θα δημιουργηθούν περισσότερες χρήσεις ιδιωτικών αυτοκινήτων. Υπάρχουν αρκετές μελέτες επίσης που αποδεικνύουν ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύγχρονο δίκτυο μεταφορών, αλλά επενδύθηκαν και τεράστιες ποσότητες στη δημιουργία υποδομών για την ε, ε, μετακίνηση ιδιωτικών οχημάτων. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική πολιτική μείωση των εκπομπών και άρα αυτά θα είναι εις βάρος της υγείας και του περιβάλλοντος. Θα ο πρόεδρος διακόπτει και ζητά από τον ε, ομιλητή να μιλήσει λίγο πιο αργά, διότι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Επειδή μου είπατε ότι έχω μένω πέντε λεπτά, τα είπα πολύ γρήγορα. Μειώθηκε λοιπόν το ωράριο των ε, μέσων μαζικής μεταφοράς, κυρίως το ωράριο του μετρό, γεγονός ε, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις και δεν θα τηρηθεί η νομοθεσία. Όλες αυτές οι πληροφορίες φυσικά είναι στη διάθεσή σας. Και τώρα, όσον αφορά την αναφορά ε, 0323 του 2011 θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να τηρούνται κάποιοι ε, ευρωπαϊκοί νόμοι ε, λαμβάνονται μέτρα για να μειωθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και να αυξηθεί η χρήση των ε, ιδιωτικών αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα με την ε, εφαρμογή ε, και την αύξηση της ρήπανση, ενώ λαμβάνονται μέτρα για να τηρηθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ε, βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης, που είναι ο βασικός παράγοντας ρήπανση. Επειδή υπάρχουν λοιπόν προβλήματα και για το Δήμο, θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία ε, λαμβάνονται δεν είναι στο ύψος της σοβαρότητας του προβλήματος. Θα θέλαμε λοιπόν να διατηρήσετε ανοιχτό το αίτημά μας ε, για να συμπεριλάβετε όλα αυτά τα νέα στοιχεία και να περιμένουμε και τη μελέτη των επιπτώσεων των μέτρων που λαμβάνονται για τα μέσα μαζικής μεταφορά στη Μαδρίτη, ε, το γεγονός ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία έχουν ε, ε, ληφθεί και επίσης να υπάρχουν στα στοιχεία της Επιτροπής Αναφοράς αξιολογήσεις για την ποιότητα του αέρα και για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα είναι διάφανα και θα είναι προς όφελος της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και να πούμε ότι δεν λαμβάνονται και κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ε, χρήσης γιοταχή αυτοκινήτων και την προώθηση της χρήσης του πεδιλάτου που είναι φυσικά πολύ λιγότερο ρηπογόνο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Συνέτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ όμως πολύ γιατί είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες για μας. Κάναμε μια συνεδρίαση τον τελευταίο καιρό με εκπροσώπους και της Ισπανικής κυβέρνησης. Το θέμα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αυτά τα οποία λέγουν οι πολίτες που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και με την υγεία στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζω στην αγγλική γλώσσα. Το θέμα είναι αρκετά ευαίσθητο και θα εκφραστώ καλύτερα στην αγγλική. Ε, σχετικά με το πρόβλημα αυτό πρέπει να το οριοθετήσουμε στο σωστό πλαίσιο. Η Ισπανία έχει πρόβλημα σχετικά με ορισμένους ρηπαντές, αλλά ε, ε αντιθέτως από ορισμένες άλλες χώρες μέλη, ε, το το ποσοστό το οποίο ε, ε, υπερβαίνει τα όρια δεν ισχύει για, την, ε, για τον αέρα. Είδαμε δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί επέτρεψαν να υπάρξει μία μείωση της ρηπάνσεως κατά 57% δημιούργησαν μία ζώνη χαμηλού, χαμηλής ρηπάνσεως. Παρ' αυτά όμως υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές ε, αλληλεπιδράσεις από γειτονικέ χώρες. Χωρίς αυτό να ισχύει για την ε, Ισπανία. Στην Ισπανία δεν υπάρχουν άλλους, άλλες ρησπάνσεις και ε, αυτού αν λάβετε υπόψη τι την νομοθεσία την κοινοτική ε, η Ισπανία έχει, ε, έχει παραβεί ε, τρεις οδηγίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα και δεν υπάρχει μία γραμμική μείωση αλλά επειδή κάπου η υπάρχει ρήπανση, μπορεί να υπάρχει διασυνοριακή επίδραση, χωρίς όμως αυτό να ισχύει για την Ισπαρία. Γι' αυτό και ζητήσαμε να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό και όσον αφορά τις άλλες λεπτομέρειες δεν θα τις σχολιάσω, άπαξ και υπάρχει ανοιχτή ε, ενέργεια επιπαραβιάσει. Ε, δεν ε, θέλουμε να αποκαλύψουμε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά ε, υπάρχει αυτή η παραβίαση και το δικαστήριο τώρα θα προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων ε, εμείς διατηρούμε ανοιχτή τη διαδικασία επί παραβάση και πέραν αυτού οι αρχές της ε, Ισπανίας ζήτησαν ε, μία επιπλέον προθεσμία εναντίον ορισμένων ρηπαντών επιπροσθέτων και αυτό αναφέρεται στην Βαρκελόνη. Έχουν ζητήσει για το θείο και για άλλους ρήπαντες ε, για την περίοδο της, ε, για την περιοχή της Μαδρίτης και όποτε υπάρχει ε, μία μία διπλή ρήπανση και υπέρβαση των φυσιολογικών τιμών ε, μπορεί να να δούμε ότι εφόσον ε, υπάρχει υψηλό επίπεδο και αζότου και ε, θείου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ε, ρήπανση από ότι την τελευταία φορά που είχε γίνει διαδικασία. Δεν θέλω εδώ να σας κουράσω αλλά ε, ε, εμείς λαμβάνουμε συχνά στοιχεία σχετικά με ένα σταθμό, όχι όμως με άλλους. Can really address the problem, because the problem there is... Και βλέπουμε ότι πολλές φορές η ρήπανση είναι ε, ε, ε, εντοπισμένη σε μία συγκεκριμένη περιοχή αλλά βέβαια ε, η λήψη μέτρων είναι στη διάκριση της εμπλεκομένης κυβερνήσεως και των τοπικών αρχών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι η αναφορά αυτή μπορεί να παραμείνει ανοιχτή αναμένοντας την απάντηση των αρμοδίων αρχών την οποία έχουμε ζητήσει διότι η Ισπανικές αρχές πρέπει να μας πούν πώς σκοπεύουν να επιλύσουν το πρόβλημα και ε, έχουν ε, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ε, ένα πρόγραμμα και μετά να το υποβάλουν προς έγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με τις παρεμβάσεις. Καταρχάς, η κυρία Ιρικογέν. Και σας παρακαλώ σύντομα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω απλώς ότι συμφωνώ με την αναφορά και θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, διότι πρόκειται για μία από τις περιοχές ε, που όπως είπατε και εσείς ε, ε, που έχουν τη μεγαλύτερη ρήπανση και μάλιστα η γειτονιά μου, το πιλάρι, είναι από αυτές που έχουν την περισσότερη ρήμα. Και όταν επιστρέφω βομβαρδίζουμε από διοξίδιο του αζήτου και όζων που μας ανησυχεί όλους. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι δίνει την ευκαιρία στι αρχέ τη Μαδρίτη να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση και να ε, δοθεί ένα τέλο σε αυτό το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει, δεν είναι πολύ δαπανηρό και μάλιστα είναι πολύ εύκολο να το θέσουμε σε εφαρμογή. Είναι αλήθεια ότι η κυρία Βοτήγια παρουσίασε ένα σχέδιο ποιότητα στο αέρα τον Απρίλιο, αλλά όπω ακούσαμε, το σχέδιο αυτό αφορά μόνο αύξηση στην τιμή των παρκόμετρων και διεύρυνση των παρκόμετρων. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα. Ε, η ομάδα σοσιαλιστών του Δήμου ζήτησε να γίνει μια έκτακτη ολομέλεια για την ποιότητα του αέρα στη Μαδρίτη. Έγινε αυτή η ολομέλεια. Το θέμα της Μαδρίτης το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι εγώ εργαζόμουν στο Δήμο, ε, στην ε, ομάδα των σοσιαλιστών του Δήμου και ε, το θέμα αυτό επαναλαμβάναμε συνεχώς και λέγαμε ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος στη ρήπανση, διότι είναι εις βάρος της υγείας του καθενός λόγω των υψηλών επιπέδων διοξιδίου του αζότου. Στο πλάι μου βρίσκεται ο σύντροφος και φίλος, ε, ο οποίος ε, θα σας πει και τι έκανε και τι έγινε στη συνεδρίαση του Μαΐου, διότι στη συνεδρίαση αυτή ξεκίνησαν και ενεργοποιήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί, 16 μέτρα, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολα ε, και συμφωνούν με αυτά όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν κάποιες περιοχές προτεραιότητας που είναι περιοχές κατοικίας και είναι πολύ εύκολο εκεί να ενταθούν οι έλεγχοι που γίνονται για την ποιότητα του αέρα. Επίσης ε, μέτρα για καθαρή ενέργεια, χρήση καθαρής ενέργειας και όλα αυτά με αιτήσει εκθέσεις. Να περιοριστεί η κυκλοφοριακή κίνηση, να αυξηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μελετηθεί η ποιότητα του αέρα στους δρόμους, να αυξηθούν οι προστατευόμενες περιοχές κατά 30%, να υπάρχει ε, διαβάθμιση στα όρια ταχύτητας ε, των αυτοκινήτων εντό της πόλης και να υπάρχουν διαφοροποίηση σε όλες τις περιοχές τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να υπάρχουν κάποιες περιοχές προτεραιότητας που είναι κατοικημένες περιοχές ε, και επίσης σε περιοχές που υπάρχουν πανεπιστήμια, ε, σχολεία και η όπερα. Όπως επίσης ε, και στην περιοχή του Κοντεντού και στην Οδό Καρέτας και σε άλλες περιοχές και να υπάρχουν ε, πεζόδρομοι, να δημιουργηθούν 10.000 θέσεις εργασία, ε, συγγνώμη, πάρκινγκ για ε, μηχανές και να αυξηθούν ε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόκειται για μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να μειωθούν τα ποσοστά διοξιδίου του αζότου και να διευκολύνουν και τη ζωή των πολιτών της ε, Μαδρίτης και να έχουμε μια πιο υγιεινή ζωή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής εδώ. Η ποιότητα του αέρα στη Μαδρίτη ε, είναι γνωστή σε όλους. Ξέρουμε όλοι τι αναπνέουμε στη Μαδρίτη. Εγώ έχω ε, Τέσσερι γιου στη Μαδρίτη και θα ήθελα ο αέρα που αναπνέουν να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτικού. Όσο καλύτερη ποιότητα έχουμε, τόσο το καλύτερο. Έχω όμω κάποιε αμφιβολίε για την αναφορά και είδα και τα έγγραφα στα οποία ε, μα επιστήσατε την προσοχή τι υπόμε... προηγούμενε ημέρε. Καταρχά, η Μαδρίτη είναι η μόνη περιοχή που αναφέρεται στην αναφορά, όταν υπάρχουν 254 περιοχέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν τηρούν τα επιτρεπόμενα όρια. Στην Μαδρίτη ε, λέγεται ότι έχουμε τα πιο αυξημένα όρια, ενώ δεν είναι αλήθεια αυτό. Γιατί επιμένουμε για τη συγκεκριμένη αναφορά όταν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι σήμερα, αλλά και γραπτός, ότι η Μαδρίτη έκανε αυτό που της αναλογούσε και ε, με ε, πράξεις απέδειξε ότι είναι αποφασισμένη να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να τηρήσει την οδηγία 08 ε, κάθετος 2004. Αναφέρονται κάποιες περιοχές ε, της Νότιας Ευρώπης, στην οποία ε, υπερβαίνονται τα όρια, διότι το κλίμα, επαναλαμβάνω, το κλίμα είναι αυτό το οποίο ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη αυτών των σωματιδίων και τη, των υπογόνων παραγόντων και μάλιστα η Μαδρίτη το κάνει πολύ καλύτερα διότι υπάρχουν κάποιες περιοχές ε, στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά. Εμείς έχουμε πολύ πιο χαμηλά ποσοστά. Αν δεν γίνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Μαδρίτη και άλλων περιοχών τη Ισπανία, δεν αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, η αναφορά αναφέρεται εδώ μόνο στη Μαδρίτη και πραγματικά αυτό εμένα μου φαίνεται περίεργο. Ολοκληρώνοντα, ε, γιατί δεν ε, προσφύγατε στη δικαιοσύνη ε, αν είστε βέβαιοι και έχετε επαρκείς αποδείξεις ότι η Μαδρίτη δεν τηρεί την 2008 ε, κάθετος 50. Ξέρετε ότι δεν προσφύγατε γιατί δεν θα περνούσε η διαδικασία αυτή. Και τέλος, να σας πω να σας πω ότι εγώ πίστευα ότι αυτή ήταν μια αναφορά για την ποιότητα του αέρα και όχι για τις τιμές των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της Μαδρίτης. Αυτά τα στοιχεία μας είπατε εδώ δεν είναι πληροφορίες, αυτές είναι απλές απόψεις οικασίας και αυτή είναι νέα αναφορά. Και κατά την άποψή μας, μια και μιλούμε για αναφορές, ε, και είπαμε ότι η πρόθεσή μας είναι να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, εντάξει να μείνει, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Άλλη είναι η ποιότητα του αέρα και άλλο είναι το τίμημα του εισιτηρίου το Μέσο μαζική ε, μεταφοράς. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω, με έχουν μπερδέψει αρκετά πράγματα. Λέτε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί ζητάτε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ποτέ δεν άκουσα να μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Εμείς θα αποφασίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει τι κάνει, αλλά γιατί μας ζητάτε εσείς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες από αυτού. Και επιπλέον μας λέτε ότι Υπάρχει δυνατότητα να δούμε τι γίνεται, περιμένουμε, είναι, ε, υπάρχει δικαστική διαδικασία να εξελίξει, τότε να περιμένουμε τι, να δούμε την απόφαση των δικαστηριών και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να συζητάμε χωρίς να αποφασιστούν τα δικαστήρια. Και επίσης λένε ότι μα ενημερώνει αναφορά. Δεν είναι αναφορά αυτή που θα μα ενημερώσει. Οι αρμόδιες αρχέ είναι αυτέ που πρέπει να μα δώσουν τα στοιχεία ε, κατόπιν αιτήματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αναφέρον δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μα δώσει τα στοιχεία. Ε, δεν ξέρω, ο Δήμο τη Μαδρίτης, η Ισπανική κυβέρνηση, κάποιο άλλο είναι αυτό ο οποίο πρέπει να διαβιβάσει τα στοιχεία. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ζητήσω είναι να κλείσει συγκεκριμένη αναφορά ή να μείνει σε κρεμότητα μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα να πω. Νομίζω ότι είναι σαφή η θέση μου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία øh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια καλή ενημερωτική απάντηση. Δεν καταλαβαίνετε τη δανεική γλώσσα. Περιμένω λοιπόν ώσπου να φορέσετε ακουστικά. Ελπίζω να συνεχίσετε λοιπόν με τον ίδιο ενθουσιασμό το θέμα το οποίο μας απασχολεί, το θέμα της Μαδρίτης. Είχα πάει μια αποστολή στη Μαδρίτη. Είδα πως ε, προσπαθούσαν να σεβαστούν το περιβάλλον και τα συμφέροντα του πολίτη. Είδα ότι υπήρχαν υπεκφυγές Προσπάθησαν ορισμένοι να μην δώσουν απαντήσεις σε σχέση ε, με κάποιους κοινοτικούς κανόνες που δεν εφαρμόζονται σωστά. Ακόμα και μικροί δρόμοι στη Μαδρίτη μετατρέπονται σε αυτοκινητοδρόμους. Και σε μία συνάντηση που είχαμε στη Μαδρίτη ε, συμμετείχαν 400 πολίτες οι οποίοι είπαν ότι για πρώτη φορά τους αντιμετώπιζαν σοβαρά. Διαπιστώσαμε επίσης ότι θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη αναδρομικών επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συμφωνήσει με αυτό, αλλά νομίζω ότι η μελέτη αυτή δεν έδωσε τις απαντήσεις που έπρεπε. Και ξαφνικά δημιουργήθηκε ένας αυτοκινητόδρομος που διέσχιζε το σύνολο σχεδόν της πόλης με πολύ υψηλά ύψη, ε, πολύ μεγάλα ύψη εκπομπών. Ευχαριστώ λοιπόν για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό σοβαρά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τη Μαδρίτη. Υπάρχουν και άλλες πόλεις στις οποίες υπάρχουν απαιτήσει για τα θέματα της μόλυνσης, οι οποίες δυστυχώς δεν, γίνονται, δεν εξυπηρετούνται σωστά στην Κοπενχάγη. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ υποδήλατο. Αυτό δείχνει ότι ζούμε σε μια πολύ σύγχρονη κοινωνία και ακόμα και οι πλουσιότερες οικονομικά τάξεις χρησιμοποιούν το ποδήλατο και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μια ολόκληρη σειρά προβλημάτων. Τα ποδήλατα κοστίζουν πολύ λιγότερο, είναι πρακτικά και κάνουν καλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ σε τέτοια θέματα έχω μια ειδική ευαισθησία. Είναι εύκολο να την έχει κανείς όταν έρχεται από εκεί που έρχομαι εγώ που έχουμε τα μέσα. Ο αναφέρον έχει το λόγο για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι το γεγονός ότι και σε άλλες προ... πόλεις έχουν περιβαλλοντικά προβλήματα, ρήπανση, οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε εμείς το πρόβλημα που καταγγέλουμε, με το πρόβλημα που καταγγέλουμε εδώ. Και γιατί η Μαδρίτη, γιατί αναφέροντας είμαστε κάτοικοι της Μαδρίτης και μας ε, πλήττει η ρήπανση της Μαδρίτης πάσχουμε καθημερινά, υπάρχουν πολύ υψηλά επίπεδα ρήπανσης και τα βλέπουμε στη Μαδρίτη, μα ανησυχούν και θέλουμε να επιληθεί. Είμαι βέβαιος ότι άλλοι πληγέντες από τη ρήπανση σε άλλες περιοχές μπορούν να, να ε, κάνουν τις δικές τους αναφορές. Ε, όσον αφορά το θέμα της τιμής των εισιτηρίων των μέσων ε, μαζικής μεταφοράς, να σας πω ότι υπάρχει άμεση σχέση της αύξησης του αριθμού των μέσων μαζικής ε, μεταφοράς ή της μείωσής τους ε, και την ε, ρήπανση. Διότι αν μειωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αυξηθεί το εισιτήριο και μειωθεί η χρήση, τότε θα χρησιμοποιούν περισσότερο όλοι το γεταχή του αυτοκίνητο. Και επομένω, όταν ε, έχουμε θέμα ρήπανση, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι μέτρα λαμβάνεται, διότι ορισμένε φορέ μένουμε στου τύπου και δεν βλέπουμε καθόλου την ουσία. Πρέπει να δούμε την ουσία και να ξέρουμε γιατί ακριβώ μιλάμε. Υπάρχουν πολλοί ισχυρισμοί που υποδεικνύουν αυτό που σας είπαμε. Ζητήσαμε ε, να έρθουν εδώ να σας το εξηγήσουν. Το σχέδιο που ανέλαβε η Μαδρίτη δεν είναι σχέδιο της μείωσης της ρήπανσης του αέρα και της βελτίωσης της ποιότητας, αλλά είναι ένα ε, σχέδιο το οποίο έχει άλλους σκοπούς. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπα και το επαναλαμβάνω είναι ότι αυτό που έκανε ο Δήμος της Μαδρίτης δεν ε, γίνεται ε, απλώς και μόνο για να ληφθούν μέτρα. Το να λέει κάποιος ε, την άποψή του για το τι συμβαίνει ε, είναι άλλο. Πρέπει να δούμε τι μας λένε τα στοιχεία. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι γίνεται μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στο Δήμο της Μαδρίτης ο Δήμος ανέλαβε, έλαβε κάποια μέτρα και υπάρχουν τα μέτρα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ, τα παρκόμετρα και ούτω καθεξής. Γιατί είναι μέτρα αυτά που δεν έχουν καμία ουσία, όπως είπατε και εσείς. Είναι μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δίνονται τέτοιες ε, απόψεις και δεν επιτρέπουμε ε, να κλείσει αυτή η αναφορά, ζητάμε να παραμείνει αναφορά για θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, είναι απλώς έκφραση προσωπικών απόψεων. Τώρα, για την προσωπική άποψη των αφέροντα για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στο Δήμο τη Μαδρίτη, νομίζω ότι αυτό δεν έχει σχέση με την αναφορά. Ο πρόεδρο, ναι, νομίζω ότι το θέμα είναι σαφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αναφέροντα για τα όσα μας είπε. Είναι στοιχεία τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Ε, μας ενδιαφέρει και η, οδηγία, εφαρμογή τη οδηγία Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της ποιότητας του αέρα που μας ανησυχεί στη Μαδρίτη. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σαφήνειά τη και για την ενημέρωση που μας έκανε. Μας είπατε ότι όντως υπάρχει παραβίαση κάποιων ανωτάτων ορίων από πλευράς ε, Μαδρίτης ε, και επομένως έχουν ξεκινήσει και σχετικές διαδικασίες επί παραβάση και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Εγώ στις 25 Μαρτίου του 2011 είχα κάνει ένα αίτημα ε, και είχα αναφερθεί σε δύο πόλεις, ε, στη Μαδρίτη όπου το διοξείδιο του αζότου είναι άνω από τα ανώτατα όρια και στη Βαρκελόνη γιατί και εκεί βρισκόμαστε στα 50 μικρογραμμάρια πάνω από το ανώτατο όριο. Ε, είναι δύο-τρει πόλει, ναι. Γιατί όμω αυτέ τι δύο πόλει, γιατί φυσικά είναι πόλη σύμβολο και αν ληφθούν μέτρα εκεί θα βοηθήσουν και άλλε ε, πόλεις. Το, ότι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες πόλεις, ε, υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να τηρείτε, την αναφέρατε κι εσείς. Και βάσει της οδηγίας αυτής θα πρέπει να ε, τηρούνται οι οριακές τιμές μέχρι το 2015. Ε, βάσει και των απόψεων λοιπόν που ακούσαμε από τις συναδέλφους θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και ελπίζω να προβορέσουμε να συνεισφέρουμε όλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κοινωνία των Πολιτών που ήταν παρούσα εδώ σήμερα, αλλά και όλοι εσείς, ώστε να μπορέσουμε να μπορέσουμε το 2015 όλες οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν καθαρό αέρα χωρίς ρήπανση. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό και περνάμε στο τελευταίο σημείο και με αυτό το τελευταίο σημείο θα ολοκληρωθεί και η σημερινή συνεδρίαση. 20. Σημείο 20. Αναφορά 0806 του 2010 του Εμμανουήλ Δομαζάκη, ελληνικής ηθαγένειας. Συγγνώμη, κυρία Μαρίνα Σταυροπούλου, λέει ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Thank you, Mr. President. Uh, we refer Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερόμαστε στην αναφορά μας της 25ης ε, Ιουνίου του 2010 και βάσει αυτής πρέπει να τονίσω ότι η προστασία του περιβάλλοντος ενδιαφέρει πάρα πολύ την εταιρεία μας και αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα του θέματος και των ερωτήσεων. Η Κρέτα φάρμ ο αναφέρον, είναι ε, μια σημαντική εταιρεία στον τομέα των τροφίμων στην Ελλάδα με ποιοτικά προϊόντα και με πολύ υψηλά υγειονομικά πρότυπα. Βάσει ε, του του, της αρχής να σκέφτεται κανείς τον κόσμο και να ε, επιδρά επί της ε, συγκεκριμένης περιοχής η η Κρέτα Φάρμα ακολουθεί τα πρότυπα της Ισπανίας και της Ιταλίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν βασιζόμαστε μόνο στο καινοτόμο δίπλωμα ευρασιτεχνίας ε, σχετικά με το λίπος των ζώων που χρησιμοποιεί αλλά χαίρεται και υπερηφανεύεται και για τις υψηλές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές που έχει ε, καθότι έχει προωθήσει την, ε, τα περιβαλλοντολογικά πρότυπα και εις την Ελλάδα και εις την Κρήτη στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οπότε από ίδια πρωτοβουλία και με υψηλό κόστος παραμένει ηγετική σε όλα τα επίπεδα όπως και στην προστασία του περιβάλλοντος καθότι ελέγχεται τακτικά από όλες τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές και έχει όλες τις αναγκαίες άδειε για τις κινήσεις της στις εγκαταστάσεις της. Σχετικά με την λεγόμενη ρήπανση Έχω σήμερα τα ε, προσκομίσει τα αποτελέσματα όλα όλων των ε, αναλύσεων που έγιναν στα ίδια ε, τα μπροστά στην, στην περιοχή, μπροστά στην εταιρεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία ρήπανση και η θάλασσα είναι κατάλληλη για κολύμπη. Η Κρέτα Φάρμ, ο αναφέρον, ε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και είναι πολύ ευαίσθητη σε θέματα περιβάλλοντος ε, που είναι προς το ίδιο συμφέρον της. Να να ε, εφαρμόζει την περιβαλλοντολογική νομοθεσία και να ενημερώνει και τον καταναλωτή. Ε, γι' αυτό και δεδομένες της σημασίας του θέματος αυτού έχουμε υποβάλει αυτή την αναφορά και απορρίπτουμε οποιαδήποτε κατηγορία για ε, παραβιάσεις της νομοθεσίας ε, για τα οποία καταγορείται. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μακάντιου, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, ε, τον Ετούντα ε, που αναφέρεται εις το περιβάλλον και όχι μόνο εις το θέμα της Κρέτα αλλά και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απήντησε σε μία γραπτή ερώτηση την οποία είχε λάβει το 2010 σχετικά με τη ρήπανση του υπεδάφους και της θάλασσας κοντά στην χειροτροφία φική μονάδα της ε, Κρέτα Φάρμ και ε, ε, η ερώτηση αυτή μας είχε παραπεμφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξού και προσεγγίσαμε τις ελληνικές αρχές για να ενημερωθούμε επί της φύσεως των αρχών ε, των εγκαταστάσεων και ε, το, εάν ε, υπάρχει ολοκληρωμένη πρόληψη εναντίον της ρήπανσης της εγκαταστάσεις αυτές. Κοιτάξαμε λοιπόν όλα τα και εξετάσαμε όλα τα περιβαλλοντολογικά θέματα και τις άδειες που έχει η εταιρεία. Οι ελληνικές αρχές μας είπαν ότι η πρώτη άδεια ε, ε, είχε χορηγηθεί το 1999, έκτοτε είχαν ε, υπάρξει ορισμένα προβλήματα με την συμμόρφωση στις άδειες αυτές. Οι εταιρείες, η εταιρεία είπε ότι υπήρχαν οι άδειες και οι βελτιώσεις είχαν γίνει και πέραν των αδειών από ίδια πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα αυτό όσον αφορά, την ενημέρωση που είχαμε προσπάθησε να διασκεδάσει την υποψία διπάνσεως και της θαλάσσης ε, εμείς δηλαδή σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε διαπιστώσει μία ρήπανση της ε, θαλάσσης λόγω της ε, εγκατάστασης αυτής της χειροτροφικής μονάδας και είδαμε το πρόγραμμα που ζήτησαν οι ελληνικές αρχές και δεν βλέπουμε να υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση εξού και περιορίζομαι σε αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, με έχουν αφήσει μόνο μου οι συνάδελφοι. Δεν έχει κανέναν εδώ. Πολύ θα ήθελα να μπορέσω να λάβω απόφαση με τους ε, συναδέλφους, κυρίως με τους Έλληνες συναδέλφους. Προτείνω λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά, να μείνει επισήμως ανοιχτή, ώστε να μπορέσει να γίνει συζήτηση με τους συναδέλφους και εν αναμονή να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για τις πληροφορίες γιατί θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να συζητήσουμε με τους συναδέλφους στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ε, παραμένει λοιπόν ανοιχτό το ζήτημα, θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για σήμερα. Πέρα τη συνεδρίαση, να σας ευχηθώ καλώ διακοπές, ε, είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό, όπου θέλετε να πάτε. Να περάσετε καλά και να γυρίσετε ανανεωμένοι για τη συνέχεια το Σεπτέμβριο.